Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, Εθνικοί Βουλευτές, κύριοι Ευρωβουλευτές και κυρίες Ευρωβουλευτές, ε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, σε το δεύτερο ήμιση της ημερίδας, υψηλού επίπεδου, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τεχνική παρατήρηση. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο σύστημα για να σημειώσουμε τα ονόματα των μελών της ε, ημερίδας που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτηση. Αλλά πρώτα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη του δεύτερου πάνελ, του δεύτερου γύρω Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μικολάη Ντογκογεύιτς, Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου, τον κύριο Άλεξ Βάιτ, πρόεδρο της κοινή Επιτροπής για τα Οικονομικά, τις Δημόσιες Δαπάνες και την ε, μεταρρύθμιση του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Εβάλο Κάλφιν, Ευρωβουλευτή και σύνησηγητή για το θέμα του, δημοσιο... του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο ε, Άλλο συνεισηγητή είναι ο κύριο Μπέγκε, ο οποίο θα λάβει το λόγο κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Και την κυρία Κρού, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σα. Χωρί άλλε καθυστερήσει, να δώσω το λόγο στον κύριο Ντογκιέβιτ. Σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι πάλι στο Κοινοβούλιο, αν και ο κύριος Δάμεν που κάθεται εδώ και εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε αυτήν την διάσκεψη καταλαβαίνει πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα για κάποιον που βρίσκεται στη θέση μας. Έχουμε τέσσερα στοιχεία στη θέση μας κυρίες και κύριοι για να βγάλουμε την Ευρώπη από την κρίση. Εφή, ε, εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών. Αυτό γίνεται με το πακέτο για τη φορολογία και τη δεσμή μέτρων ε, που λέγεται six Επίσης, καλύτερο ευρωπαϊκό διακανονισμό του οικονομικού τομέα και αυτό είναι ήδη που κάτι που συμβαίνει. Περισσότερη αλληλεγγύη, επίδειξη αλληλεγγύης, ιδίω ενό τείχου προστασία για το ευρώ. Και το τέταρτο στοιχείο, σε αυτό θέλω να σταθώ σήμερα, είναι η ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την ανεργία, τις, τα σημάδια ύφεση, το πρόβλημα της αντιευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, και βεβαίως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχυθεί με, παρά την κρίση στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που να είναι ένα πρακτικό εργαλείο στη Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει τις προοπτικές για ανάπτυξη στο μέλλον και για θέσεις εργασίας βεβαίως. Με μια απλή ματιά στο τι λένε οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγηση, όπω η Standard Poor's του τελευταίου μήνε, και δούμε πώ βαθμολογούν ε, τη, πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλέ υποβαθμίσει. Ακριβώ Ακριβώς δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση που, να, που έχουν προκαλέσει τα μέτρα τη λιτότητα. Νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα χρειάζεται πειθαρχία και λιτότητα, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, ε, τελμάτωση και την, τον αποπληθωρισμό που θα μας οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύκλο. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε, θα πρέπει να δούμε μάλλον το δημοσιονομικό πολιτές πλαίσιο σε ένα επενδυτικό εργαλείο. Κάτι που θα μας επιτρέψει να τονώσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά επίσης. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα επενδυτικό και βεβαίω ε, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τι κρατικέ επενδύσει. Στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει λάβει υπόψη το ισχύον ε, οικονομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Πριν κάποια χρόνια, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό οδυναμούσε με το 1,18 του ευρωπαϊκού εγχώριου, εγχώριου προϊόντος. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 1,12%, και στο μέλλον θα είναι 1,05%. Αυτό επηρεάζει όλε τις μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Εάν δείτε τα στοιχεία για τα τελευταία 10 χρόνια, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό μεταξύ του 2000 και του 2010 έχει αυξηθεί κατά 37,5%. Εν τω μεταξύ, 12 νέα κράτη-μέλη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη νέα συνθήκη με νέε αρμοδιότητε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και νέε κοινωνικέ, οικονομικέ και πολιτικέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα, εάν δούμε του εθνικού προπολογισμού, στην περίοδο αυτή 2000-2010 έχουν αυξηθεί κατά 62%. Πέρυσι μόνον μια χούφτα κράτη-μέλη περιέκοψαν τις δαπάνες τους. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε με κάθε σοβαρότητα ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν μπορεί να γίνει από διοπομπαίο τράγο για τι ε, ανεύθυνε φορολογικέ και δημοσιονομικέ πολιτικέ σε εθνικό επίπεδο. Επίση, λίγα λόγια <clears throat> για την πολιτική συνοχή. Στην Πολωνία αυτό γίνεται, αυτή η πολιτική γίνεται αντιληπτή ω μια πολιτική επενδύσεων που έχει επιτρέψει ω τώρα στην Πολωνία να κάνει ένα άλμα το 40% του μέσου όρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 στο 65% μόλι πέρσι. Βεβαίω, η συνοχή δεν μπορεί να είναι μια θεωρητική μόνο πολιτική. Είναι πολιτική που αφορά και την ενιαία αγορά ταυτόχρονα. Και η νέα αγορά είναι εκείνη, εκείνη που προσφέρει τα περισσότερα ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτε. Είναι ένα πυλώνα τη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η δαπάνε των Ευρωπαίων βεβαίω στηρίζουν τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι επενδύσει, στην ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο σημαίνει ότι έτσι θα επενδύσουμε στην ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Επίση, πρέπει η ανταγωνιστικότητα να φανεί και σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά προϋπόθεση για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας είναι και η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Άρα η ανταγωνιστικότητα και η αλληλεγγύη πάνε χέρι-χέρι. Δεν είναι αντίπαλοι. Βεβαίως, συχνά αναρωτιόμαστε το κατά πόσον τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στι διάφορε οικονομίε έχουν να κάνουν και με την πολιτική συνοχή. Αυτή η συζήτηση πολύ συχνά οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο ευθύνεται η έλλειψη ελέγχου μέτρων ε, εξονυχιστικού ελέγχου σε επίπεδο ευρωζώνη και δεν φταίνε οι συνέπειε συγκεκριμένων πολιτικών με συγκεκριμένα μέτρα. Δεν οδήγησαν αυτά στη σημερινή κρίση του δημοσίου χρέους και την κρίση εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη. Δεν μπορεί να φταίει μια ευρωπαϊκή πολιτική ή κάποια άλλη. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την ανάγκη πολιτική συνοχή να γίνει αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και ανάλογη προ το κόστο που επιβάλλει. Αλλά το ίδιο και για άλλε πολιτικέ, μεταξύ των οποίων και η αγροτική προφανώ. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα εξή στοιχεία προκειμένου το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να γίνει μια σκόπιμη απάντηση στις σημερινές προκλήσεις. Να χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό ως επενδυτικό εργαλείο. Να τον αξιοποιήσουμε ως ένα μοχλό για την ανάπτυξη. Για να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας και ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα οικονομικά δεινά παρά να θεωρείται πηγή τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Mr. White, for the Irish Parliament. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, ε, κύριε Επίτροπε, ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σήμερα το απόγευμα σε αυτήν την σημαντική συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ε, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μεν προϋπολογισμός, είναι όμως και ένα πλαίσιο. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να κάνουμε ένα βήμα πίσω, ε, να ε, ξεφύγουμε λίγο από τις διαπραγματεύσεις για τις ε, επιμέρους γραμμές του προϋπολογισμού και δεν υποτιμώ τη σημασία τους, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τα μεγάλα στρατηγικά θέματα που θέλουμε να απαντηθούν σε αυτήν τη διαδικασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε στην αρχή της συζήτησης αυτής πόσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε, πόσο φιλόδοξοι είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε κατά τον προγραμματισμό της επόμενης φάσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι με πολλούς τρόπους ο προπολογισμός είναι η Ένωση. Στα μάτια των ε, πολιτών, σε μεγάλο βαθμό, αυτά που κάνει η Ένωση, αυτά που μπορεί να πετύχει, ε, τα προγράμματα που χρηματοδοτεί, όλα αυτά γίνονται μέσω του προϋπολογισμού και γι' αυτό αυτά ουσιαστικά αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλούς τρόπους. Ας κάνουμε λοιπόν ένα βήμα πίσω και ας δούμε τα ε, μεγάλα στρατηγικά θέματα και τις μεγάλες στρατηγικές ευκαιρίες που έχουμε. Άκουσα αυτό που είπε ο Υπουργός ε, και άλλοι που θεωρούν ότι το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το μέσο ε, με το οποίο μπορούμε να πετύχουμε ε, το πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό σημείο κίνησης, διότι οι εμπειρίες στη χώρα μου, όχι όμως μόνο εκεί, είναι ότι έχουμε μια συνεχιζόμενη συζήτηση για τη λιτότητα και την ανάγκη για λιτότητα, την οποία νομίζω ότι πολλοί κόσμος ε, δέχεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Πάρα πολύ λίγοι όμως, ε, πιστεύω, ελπίζω, ε, θα μπο... πιστεύουν ότι η λιτότητα από μόνη της θα μπορέσει να αποτελέσει λύση για την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια εύρωστη πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και καταλαβαίνω αυτούς που θέλουν ε, να περιγράψουν τη διαδικασία αυτή και τη συμφωνία που θα προκύψει από αυτήν ως ε, προϋπολογισμό επένδυσης. Νομίζω ότι αυτή είναι σωστή ετικέτα. Τέτοιος θα πρέπει να είναι ο προπολογισμό επενδυτικό. Και του επόμενου μήνε ε, στην Ιρλανδία ε, θα συζητήσουμε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Πολλοί κόσμοι λέει ότι υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά τη λιτότητα. Μπορεί να μα αρέσει, αλλά καταλαβαίνουμε τι είναι. Καταλαβαίνουμε τη λογική πίσω από αυτήν και την ανάγκη ε, για λιτότητα. Αλλά είναι πιο ασαφές το τι είναι οι συνοδευτικές πολιτικές για την ανάπτυξη και ε, την απασχόληση. Μιλάμε πολύ για αυτά, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε μια μάρκα πάνω σε αυτό, όπως γίνεται στις διαφημίσεις. Ε, δεν έχουμε καταφέρει να τους δείξουμε τι είναι η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ε, αυτή λοιπόν είναι η ευκαιρία που έχουμε να καταλήξουμε σε έναν προϋπολογισμό ο οποίος ε, θα ανταποκριθεί στην σημαντική πρόκληση ε, της ανάγκης για ανάπτυξη και επενδύσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και δεν θέλω να επιμείνω στη δική μου χώρα. Να πω μόνο αυτό, ότι όσον αφορά τις εμπειρίες μας ε, ως ε, ε, ενθουσιώδης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ καλές οι εμπειρίες μας με, την, ε, με τα περιφερειακά ταμεία, τα, το Ταμείο Συνοχής, τα διαρθρωτικά ταμεία. Ήταν εξαιρετικές οι εμπειρίες που είχαμε. Και από πού ήρθε το κίνητρο τα τελευταία 30 χρόνια στην ανάπτυξη της Ιρλανδικής οικονομίας Πού είδαμε ε, παρέμβαση από πλευράς του κράτους. Από την Ευρώπη ήρθε αυτό. Και τώρα έχουμε μια σημαντική ευκαιρία και ανάγκη στη νέα εποχή μας για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, παράσχει αυτό το ζωτικό στοιχείο, έναν προϋπολογισμό επενδύσεων για να μπορέσουμε ε, να περάσουμε στην ανάκαμψη. Ε, αυτή η διαδικασία ελπίζω ότι θα διασαφηνίσει τι εννοούμε όταν λέμε μια ε, πολιτική για ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αυτή την εβδομάδα στην Κοπεχάγη ε, κάποιος στο κοινό σε μια διάσκεψη μας ρώτησε για τον Λόρδο Κέιν και ο ε, Επίτροπος Λεβαντόφσκι είπε ότι ο κεινσιανισμός δεν ε, είναι ε, δυνατό να εφαρμοστεί σε μεμονωμένες χώρες. Υπήρχε κάποια φράση για τον σοσιαλισμό σε μία χώρα. το ίδιο, κάτι παρόμοιο ισχύει για τον κενσιανισμό. Πρέπει να το έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τους ανθρώπους, θέλουμε όμως να ανανεώσουμε και το όραμα των ανθρώπων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι ε, η ευκαιρία που έχουμε. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια να ασχολείται με δημοσιονομικές περικοπές ε, να πατάει το φρένο. Ε, θα πρέπει, αφού ζητάμε τους, τις ψήφους των ανθρώπων θα πρέπει να δείξουμε επιτεύγματα, ευκαιρίες για τους νέους και να μην ε, φρενάρουμε ε, όσον αφορά τις μελλοντικές τους δυνατότητες. Και βλέποντας τις προτάσεις της Κομισιόν, ε, μπορεί κανείς να συζητήσει τα, τα επιμέρους στοιχεία, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις προτάσεις στον τομέα ε, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Εάν εφαρμοστούν τα στοιχεία αυτά και δεν θέλω να αρχίσω να μπαίνω σε νούμερο όσον αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού, εάν εφαρμοστούν όμως αυτά, θα μπορέσουμε να ε, στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, ε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για το μέλλον όσον αφορά την δημογραφική εξέλιξη και την περίθαλψη. Ε, θα μπορέσουμε έτσι να ε, ε, δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους της Ευρώπης, όχι μόνο σε αυτούς που θα αποφεληθούν από τις πρόοδους αυτές, αλλά και αυτούς που θα έχουν θέσεις απασχόλησης για τους εαυτούς τους και για τις οικογένειές τους για το μέλλον. Ελπίζω πραγματικό λοιπόν ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι προϋπολογισμός επενδύσεων και προβλέπω σε μια, προβλέπω σε μια καλή συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κάλφιν, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, παρόλο που έχουμε διαφορετικές απόψει για πολλά θέματα. Είναι ωστόσο σημαντικό να ακούμε τα επιχειρήματα τη άλλη πλευρά. Και θα ξεκινήσω και στη συνέχεια θα ζητήσω από τον συνάδελφο κ. Μέργερ να συνοψίσει γιατί δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε και είναι μέλος του Κοινοβουλίου που είναι ιδιαίτερος πεπειραμένος σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Όταν μιλούμε και ακούμε τα επιχειρήματα ακολουθούν μια ξεκάθαρη γραμμή. Υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση απαιτεί δημοσιονομική λιτότητα, περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζεται χωρίς να συζητιέται. Και τώρα θα ήθελα να επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες για να δούμε κατά πόσο ισχύει επακριβώς. Ποιο είναι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια δεδομένα γιατί δεν έχουμε πολύ συχνά αρκετές ε, πληροφορίε. Καταρχήν, διαφέρει πάρα πολύ από τους εθνικούς προπολογισμού. Το πρώτο χαρακτηριστικό ότι είναι 44 φορές χαμηλότερο από τους εθνικούς προπολογισμού για τους φορολογούμενους το 2010 η εισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ισοδυναμούσε με ένα φλιτζάνι καφέ αναμέρα. Ε, 75 ε, ε, cents τη μέρα. Εάν συγκρίνουμε πόσοι εργάτες εργάζονται σε διάφορες χώρες μέλη για να πληρώσουν τους φόρους τους μέχρι το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι κλπ. Μέχρι τις 4 Ιανουαρίου εργάζονται οι εργαζόμενοι για να πληρώσουν τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό. Εάν το συγκρίνουμε με το επίπεδο των εθνικών προπολογισμών και πούμε να γίνουν περικοπές, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι κατά 44 φορές χαμηλότερος από τους εθνικούς προπολογισμού. Δεύτερον, πρόκειται για ένα προπολογισμό επενδύσεων. Αυτό το είπαμε ήδη. 94% του ευρωπαϊκού προπολογισμού επιστρέφει στις χώρες μέλη. Μόνο 6% χρησιμοποιείται για διοικητικές δαπάνες. Και για δείξτε μου ένα τέτοιο εθνικό προπολογισμό που φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται για ένα διοικητικό άχθος που φορτώνεται στις πλάτες των πολιτών. Τώρα, όταν μιλάμε για εξηγήνιση του προπολογισμού, σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εξυγίανση του προπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν εμφανίζει ελλείμματα. Βεβαίω θα πρέπει να αλλάξει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό είναι γεγονό. Εάν δούμε την πρόταση τη Επιτροπή, ε, δείχνει μία μείωση. Με όρου αποτελεσματικότητα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σχέση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μια καλύτερη ισορροπία. Ναι, εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ε, και υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω περικοπές ε, των ε, δαπανών. Στην ουσία, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις που γίνονται μέσω του προπολογισμού αντιπροσωπεύουν εξοικονομήσεις από τους εθνικούς προπολογισμούς επιφέρει δηλαδή επιπλέον οικονομία σε εθνικού προπολογισμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση, για, το, για την εκπλήρωση των κριτηρίων του Sixth Pack κλπ. Ορισμένοι συνάδελφοι σήμερα το πρωί μίλησαν για κάποιε ενδείξει που προέρχονται από την πλευρά των ψηφοφόρων. Βεβαίω ε, ακούμε τη φωνή των ψηφοφόρων. Οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια ψηφίζουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένουν μια πολιτική με συνοχή. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια πάλι μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει περισσότερα χρήματα. Όχι, έχουμε του ίδιου, το ίδιο εκλογικό σώμα. Και όταν τα Εθνικά Κοινοβούλια επικύρωσαν τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, αυτό ακριβώς έγινε. Οι ψηφοφόροι ε, δεν έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο πράγματι εννοούσαν όλα αυτά, κατά πόσο ήθελαν να εκπληρώσουν τους στόχους, αλλά ήθελαν να κάνουν μεγαλοσχήμονες εξαγγελίες από τη μία και από την άλλη να προβαίνουν σε συνεχείς περικοπές. Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο στοιχεία όσον αφορά την πολιτική συνοχή, γιατί ε, ε, έχει γίνει αντικείμενο πολλά συζητήσεων. Με τις μεταξύ του 2002 και 2006 υπάρχει μία αύξηση κατά 0,7% του ΑΕΠ το 2009 και θα πάει στο 0,4% λόγω της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη των 25 το 2020. Θέλουμε μια τέτοια αύξηση, μιλούμε για αύξηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής ή θέλουμε να έχουμε ένα, μια ε, πολιτική η οποία αυξάνει το ΑΕΠ ενώ η οικονομική δύναμη των χωρών μελών μειώνεται. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να έχουμε και το ξεκινήσαμε ήδη, να έχουμε μια πολύ πλατιά συζήτηση με το Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο για την αύξηση, για την μεγέθυνση και για τις θέσεις απασχόλησης, ένα εργαλείο σύγκλησης και όσον αφορά τη διαδικασία θα πρέπει να είναι πολύ πιο ευέλικτος με τον ίδιο τρόπο που γίνονται πιο ευέλικτοι οι εθνικοί προπολογισμοί σε, περιπτω... σε περιόδους λιτότητας. Τώρα, αυτό που οι Ευρωπαίοι προτείνουν είναι μία μείωση του ευρωπαϊκού προπολογισμού με σχετικού όρους. Οι πληρωμές ήταν 1,8%. Τώρα με την πρόταση ε, της Επιτροπής πάνε 0,95%. Άρα έχουμε 20% μείωση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ταυτόχρονα, εάν δούμε τους εθνικούς προπολογισμούς, τότε θα δούμε μια τεράστια αύξηση των εθνικών προπολογισμών. Το 2011 23 από τις 27 εθνικούς προπολογισμούς αυξάνουν. Το 12 24 από τους 27 προϋπολογισμούς αυξάνονται και συνεχίζουμε να μιλούμε για μια μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε και μετατοπίζουμε εξουσίες από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο. Αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα δεν μπορούν να εκπληρώνονται ε, σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, μετά την επικύρωση της συνθήκης Λισαβόνας και υπόθηκε ήδη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα κρίση. Η κρίση είναι ιδιαίτερως έντονη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να εκπληρώσουμε τους πολιτικούς ε, στόχους. Δεν θέλουμε να εκπληρώσουμε τους πολιτικούς στόχους των εθνικών κυβερνήσεων, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε μια συνέπεια. Κυρία Κρούς, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά μας εμπνέει να ξεκινάμε από το σχόλιο το, περί των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει υπόψη της το θέμα αυτό. Είναι ένα από τα ζητήματα όπου εγώ μόνο τις ευλογίες μου μπορώ να δώσω και υπήρξα πολύ προσεκτική ώστε να ακολουθήσω αυτό το ίδιο πνεύμα ε, τις ε, παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια ζητήματα εφήγησαν ήδη. Για μένα είναι δύο τα βασικά μήνυματα τα οποία πρέπει να αντλήσουμε από την κρίση. Δύο διδάγματα. Ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ανάπτυξη. Πρέπει να την ενθαρρύνουμε, να την υποδαβλίσουμε, να την ε, προσελκύσουμε και να επενδύσουμε σε αυτήν. Το δεύτερο είναι ότι οι οικονομίες μας είναι αλληλένδετες, τελείως αλληλένδετες. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Το ξέρουμε όταν συζητήσαμε και για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Προφανώς πρόκειται για σχέσεις αλληλεξάρτησης. Όταν τα πράγματα όμως πηγαίνουν άσχημα, στην περίπτωση της αλληλεξάρτησης, προφανώς όλοι ε, αισθάνονται τις ίδιες συνέπειες. Δεν είναι θετικό αυτό και πρέπει να το έχουμε υπόψη. Όμως, εάν συνεργαστούμε στενά σε περιοχές ε, κοινών ενδιαφέροντος, υπάρχουν τέτοιοι τομείς, τότε μπορεί να αισθανθούμε και τα ωφέλη. Και τότε μπορούμε να μιλάμε για οικονομίες κλίμακας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας δύναμη και να γίνουμε οικονομικός πρωταγωνιστής ε, στην ε, γη, αν μπορώ να το πω αυτό. Και θα μπορούσαμε να έχουμε και θετικές παράπλευρες συνέπειες η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει ηγετική δύναμη στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτό πρέπει να μας εμπνέει. Δεν είναι απλή επιλογή βεβαίως, αλλά θα πρέπει να μας ε, εμφυσίσει θάρρος. Η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, γιατί μιλούσαμε για ένα σήμα εδώ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωση, σφραγίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον όρο πιο ε, ελκυστικό από την Ευρώπη του 2020, αλλά αυτό το αποφασίσετε εσείς, Πρόεδρε. Ε, είστε πιο αρμόδιος από μένα για να το αποφασίσετε κάτι τέτοιο. Μπορεί να βρείτε κάποιο καλύτερο όρο. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική για το 2020 είναι το δικό μας όραμα για την οικονομία. Και αυτό το χρειαζόμαστε για την επόμενη δεκαετία. Είναι σαφές. Τώρα, το σημαντικότερο είναι πώ θα πετύχουμε τα αποτελέσματά μα. Τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε, ακόμη και σε καιρού λιτότητα, όπω ήδη αναφέρθηκε, η λύση προφανώ δεν είναι να διακόψουμε τι επενδύσει. Αυτό θα ήταν απολύτω ανόητο. Θα έλεγα το ακριβώ αντίθετο ισχύει. Σε πολλέ περιπτώσει, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα, είναι ένα μέσο στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε για το μέλλον, ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα από το δικό μου χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων, το οποίο είναι οριζόντιο. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν και έχουν λόγο και είμαστε και πολύ κοντά στι ανάγκε του καταναλωτή και του πολίτε. Τρόπον τεινά. Εσείς μιλήσατε για το δυναμικό μας, του ενδυνάμει ψηφοφόρου μας μάλλον. Όλοι ε, έχουν, ε, επηρεάζονται από το χαρτοφυλάκιο αυτό. Ήδη σήμερα η ψηφιακή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερη από του Βελγίου και μεγαλώνει ταχύτερα από ό,τι τη Κίνας οι νέε λύσει, οι καινοτόμε λύσεις, από τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι το smartphone μπορεί να έχετε στην τσέπη σα, όλα αυτά είναι φαλτήρια για την καινοτομία. Νέε υπηρεσίες, νέα προϊόντα και νέε εφαρμογές. Και δεν είναι μόνο για σκοπούς ψυχαγωγία, ούτε για... Ακόμη και αν κάποιοι το χρησιμοποιούν για σκοπούς διασκέδαση. Αυτό είναι θέμα του καθενό. Όχι, χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά και για κοινωνικού σκοπού. Το υπολογιστικό νέφο θα δώσει στι στις ε, μικρέ επιχειρήσει τα ευέλικτα εργαλεία για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικέ. Ακόμη και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να μειώσουν τα, τις δαπάνες των κυβερνήσεων. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική μου σταδιοδρομία, κύριε και κύριοι, που φίλοι μου, υπουργοί οικονομικών, γνωρίζουν ότι με την ψηφιακή αυτή προσέγγιση, μιλώντας για την ηλεκτρονική υγεία, μιλώντας για τη γύρανση του πληθυσμού, μπορεί τελικά να έχουμε στα χέρια μας ένα τεράστιο όπλο για να μειώσουμε τα πάνω στον προπολογισμό Συνολικά όλα αυτά τα μέσα της καινοτομίας μπορεί να μας επιτρέψουν να κάνουμε ένα άλμα στην παραγωγικότητα, στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μια από τι πιο ευχάριστε εμπειρίε που είχα ήταν ε, στα παρασκήνια του Σώματος των Επιτρόπων, όταν μιλούσαμε για την ανάπτυξη και την οικονομία και τις θέσεις εργασίας, όπου ο πρόεδρος αναγκαστικά μας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, τα οποία δυστυχώς είναι καταφληπτικά, είναι όλα αρνητικά. Όμως στον τομέα ICT, στην τομέα της πληροφορικής, εδώ είναι ο μόνος τομέας που βλέπουμε ότι τα πάντα είναι σε τάση, έχουν τάση αυξητική, θετική και υψώνονται. Έτσι λοιπόν, το να μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας, για ανάπτυξη τα ερχόμενα ε, χρόνια είναι πολύ θετικό. 7.000 θέσει εργασία θα καλυφθούν τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Το γνωρίζουμε. Απλώ θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και εμεί και οι πολίτε και οι νεότερε γενιέ. Είναι απέσια τα ποσοστά ανεργία των νέων, οπότε θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια από τα κενά που υπάρχουν. Ήδη σήμερα ε, η κίνηση στο διαδίκτυο έχει διπλασιαστεί και διπλασιάζεται κάθε δύο με τρία χρόνια. Όλο το περιεχόμενο αυτό, το νέο υλικό, είτε μιλάμε για ταινίε online, επιγραμμικέ ταινίε, είτε για ε, προβολές ταινιών ε, στο διαδίκτυο, όλα αυτά λειτουργούν πλέον ευρυζωνικά. Το να στηρίξουμε λοιπόν την ανάπτυξη αυτή, αυτές τις εξελίξεις, χρειαζόμαστε νέες υποδομές, όχι αυτές που έχουν μια, την ηλικία τουλάχιστον 10 ετών, αν δεν επενδύσουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, σε λίγα χρόνια η έλλειψη δυνατοτήτων στο ε, διαδίκτυο θα αποστραγγίξουν όλο αυτό το δυναμικό, θα στραγγαλίσουν την καινοτομία. Όλες αυτές οι νέες εφαρμογές, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να διασυνδεθούν με την οικονομική ανάπτυξη, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν τώρα δεν προετοιμαστούμε, εάν δεν προσφέρουμε μόνο νέες υπηρεσίες, αλλά και περιεχόμενο, δεν θα έχουμε τους σωστούς διάβλους, την υποδομή και θα χάσουμε πολλές ευκαιρίε. Η έλλειψη δυνατοτήτων λοιπόν στο διαδίκτυο θα φραγκαλίσει αυτό το δυναμικό. Εάν με ρωτήσει κανεί ποια είναι η μεγαλύτερη μου μέρη, είναι ακριβώς αυτή η πιθανότητα. Το γνωρίζουμε, ξέρουμε τι οφείλουμε να κάνουμε και να, μπορεί να μην κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Εδώ πρέπει να αντισταθούμε. Αλλά εάν επενδύσουμε, και αυτό είναι η θετική σκοπιά, θα δούμε τα ωφέλη. 10 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρυζωνική δίσδυση σημαίνει μία με μία μισή ποσοστία μονάδα αύξηση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Είναι καλές ειδήσει για τις σημερινές μέρες, για τη σημερινή περίοδο. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε στο ευρυζωνικό διαδίκτυο. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως δεν αρκούν για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι όμως ζωτική σημασία να μειώσουμε το ποσοστό κινδύνου αυτών των προγραμμάτων και να μοχλεύσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις που χρειαζόμαστε για να γίνουμε μια ήπειρος ανταγωνιστικά διασυνδεδεμένη. Με αυτό το είδος ευφυούς καινοτόμου ε, χρηματοδότησης, το μέσω διευκόλυνση διασυνδέοντας την Ευρώπη θα μα δώσει πολλέ καλέ λύσει για το ευρυζωνικό διαδίκτυο. Τώρα, ε, για τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για το Connecting Europe 9,2 δις ευρώ θα πρέπει να βρούμε ένα ευφιέστερο σύστημα χρηματοδότησης με μόχλευση με την συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να φτάσουμε κατά 200 δι ευρώ. Τότε θα μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Τότε θα είμαστε ξύπνοι. Μπορεί να ε, έχουμε πραγματική διασύνδεση διακρατικά, ακόμη και με περιοχέ τη επέθρου. τετοιε Τέτοιε λύσει χρειαζόμαστε. Ένα άλλο η E-government, ηλεκτρονική κυβέρνηση. Εδώ μπορούμε να έχουμε διάδραση μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων με τρόπο και απλό και φτηνό. Όμως σε μια ενιαία αγορά τα συστήματα θα έπρεπε να λειτουργούν και εκτός των συνόρων. Θα... Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντική η διευκόλυνση για την διασύνδεση της Ευρώπης. Εάν λάβουμε τις σωστές αποφάσεις και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τότε μπορούμε να τα πάμε καλά. Ένα άλλο παράδειγμα Εάν θέλουμε να τονώσουμε την παραγωγικότητα του μέλλοντος, πρέπει να δώσουμε όθηση στην καινοτομία και την έρευνα. Ήδη οι νέες τεχνολογίες με τις ε, μελέτες που γίνονται μπορούν να αναπτύξουν την τεχνολογία μας και αυτό μπορεί να γίνει από τα νανοηλεκτρονικά με τις, υψηλής, με τις ε, τελευταίες ε, υπολογιστές με το διαδίκτυο του μέλλοντος. Εάν αυτά τα ακολουθήσουμε ως πηξίδα για το μέλλον, θα καταλάβουμε τελικά τι μπορεί όλα αυτά να εκπροσωπούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο καιρό επένδυσε 120 εκατομμύρια ευρώ στην τεχνολογία και αυτό για ερευνητικά προγράμματα της Επιτροπής και μόνον. Έτσι καταλήξαμε σήμερα να έχουμε την αγορά 3G για τα κινητά τηλέφωνα όχι μόνο αξίζει 250 δις αυτή η αγορά αυτή τη στιγμή, αλλά σκεφτείτε τι δυνατότητες έδωσε. Όχι μόνο εφαρμογές που έδωσαν δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και εργαλεία που διευκολύνουν τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, των πολιτών. Τέτοιου είδου απόσβαση των επενδύσεων μπορούμε να λάβουμε από την εύρωστη έρευνα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Horizon 2020, τον ορίζοντα του 2020. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του τι εννοούμε με το μελλοντικό ε, πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορούμε να έχουμε πραγματική οικονομική αναγέννηση στην Ευρώπη. Και αυτό το χρειαζόμαστε παγκοσμίω. Με καινοτόμα προπολογισμό που να ανταποκρίνεται στι σημερινέ προκλήσει και να δημιουργεί ευκαιρίε για το αύριο. Εδώ υπάρχουν πραγματικέ ευκαιρίε. Θα πρέπει όμω να έχουμε σωστή στοχοθεσία. Έχουμε τα εργαλεία που θα μα το επιτρέπουν αυτό. Πρέπει να αδράξουμε τι πραγματικέ ευκαιρίες που υπάρχουν. Αυτό είναι το σλόγγαν μα. Θα πρέπει να μας βοηθήσετε, να εξηγήσετε κι εσεί, στο δικό σα περιβάλλον, στο δικό σα κύκλο, ότι αν επενδύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επενδύσουμε σε ένα πραγματικό μέλλον. Σα ευχαριστούμε κυρία Κρούς και τώρα να δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες που έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Έχουμε αρκετού ε, που ενδιαφέρονται να πάρουν το λόγο. Αλλά θα πρέπει να παραμένετε στα δύο λεπτά περίπου ανά ομιλητή. Πρώτος, ο κύριος Μέλουνας από την Λιθουανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Να πω καταρχήν ότι δεν μπορώ να φανταστώ καμία ευρωπαϊκή πολιτική που να οδηγεί σε ε, καλύτερο μέλλον εάν δεν έχει έναν αξιόπιστο και σοβαρό προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό για επενδύσεις που να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες ε, δεκαετίες. Οι κοινέ ε, πολιτικές γεωργίας και συνοχή εισήχθησαν πριν κάποιες δεκαετίες και έχουν οδηγήσει σε πολλές αλλαγέ γύρω μας τα τελευταία χρόνια. Πρόκληση αποτελεί η σοβαρή οικονομική κρίση, τα μέτρα λιτότητας λόγω του ανταγωνισμού την ε, αλλαγή του κλίματος κτλ. Αλλά ε, στόχος είναι να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Ποτέ δεν χρειαζόμασταν περισσότερο τέτοιες ε, πολιτικές, την, πολιτική, της κοινής, την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Να σας πω μια ιστορία επιτυχίας από τη χώρα μου, την Λιθουανία. Στα νότια της Λιθουανίας υπάρχει μια μικρή πόλη, η Τρισκονίσκε, που ήταν ε, πολύ γνωστό θέρετρο ε, πριν κάποια χρόνια. Το 2013, ε, το 2003 τα έσοδα εκεί ήταν υψηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη η χώρα, ε, αλλά ε, μετά η ελκυστικότητα του τόπου αυτού χάθηκε. Ε, χάρη όμως στις επενδύσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, εννέα χρόνια μετά έχει εξυγχρονιστεί η υποδομή της πόλης, έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις απασχόλησης και έχει ξαναγίνει ελκυστικό θέρετρο, για, ε, θέρετρο, που προσελκύει όχι μόνο τουρίστες, αλλά και τουρίστες από γειτονικές χώρες. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Υπάρχουν όμως χιλιάδες ιστορίες επιτυχίας σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι κοινέ πολιτικές όπως η πολιτική συνοχή και η κοινή γεωργική πολιτική έχουν ε, αποτελέσει πηγή επενδύσεων και έχουν ε, οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρξει ε, εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ισχυρή εσωτερική συνοχή. Και κυρίες και κύριοι να κλείσω λέγοντας ότι το μέλλον μας εξαρτάται και από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις, να καταπολεμήσουμε την ε, κρίση, να ε, καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος ε, κλπ. Εάν θέλουμε να πετύχουμε θα πρέπει να έχουμε ισχυρή εμπιστοσύνη στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες φέρνουν αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ πολύ κύριο Μελούνας. Ε, η Ουγγαρέζη Υπουργό ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Τρει γενικέ παρατηρήσει ε, θα ήθελα να κάνω. Θα μακρηγορήσω λίγο, αλλά όχι πάνω από δύο λεπτά. όταν ασχολούμαστε με το θέμα του πολιετού οικονομικού πλαισίου, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι καθορίζουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχου μα και δεν φτιάχνουμε έναν προπολογισμό λιτότητα για σύντομο χρονικό διάστημα. Η η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει αυξήσει τι αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ σωστά είπε ο Προεδρο. Δεν ε, μπορεί να απαιτηθεί από εμά να αναλάβουμε αυτά τα καθήκοντα, εάν δεν υπάρχει επαρκή ε, χρηματοδότηση. Όλοι συμφωνούμε ότι το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει του στόχου τη ε, πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρί βελτίωση τη εσωτερική συνοχή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να πω λίγο, λίγα λόγια παραπάνω για τις ε, παραδοσιακές πολιτικές, την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής, ε, διότι ε, είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις πολιτικές αυτές ως ισχυρές κοινωνικές πολιτικές ακόμα και στο επόμενο πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, να θέσει ανώτατο όριο 2,5% ε, του ΑΕΠ όσον αφορά τα, τη χρηματοδότηση συνοχής για τα κράτη είναι άδικη. Είναι ιδιαίτερα άδικη η πολιτική αυτή για τα, τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Αποτελεί αυτό το βασικό μας εργαλείο για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική συνοχής βοηθάει οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχέ ε, να μπορέσουν να φτάσουν το επίπεδο των άλλων. Ε, δεν ε, μα ενδιαφέρουν μόνο αυτές όμως περιοχές, ε, συγγνώμη, εταιρείες των πιο αναπτυγμένων κρατών μελών σίγουρα υποφελούνται από, την, από τα προγράμματα αυτά. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι κάθε ευρώ συνοχής που επενδύεται δημιουργεί 61 λεπτά κέρδος για ε, τις άλλες χώρες. Με άλλα, λεπτά, με άλλα λόγια, τα 61% των ε, των ε, χρημάτων που επενδύονται στις μη αναπτυγμένες περιοχές καταλήγουν στα χέρια εταιριών από μη μειονεκτικές περιοχές. Με άλλα λόγια, επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουν περισσότερα, εποφελούνται από ε, τα Ταμεία Συνοχής στην εποχή μας όπου μας έχουν εξαντληθεί τα κεντζιανά μέσα ε, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο στόχος της σημερινής συζήτησης είναι να εντοπιστεί να καθοριστεί ο λόγος ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ως ε, μέσο για την ανάπτυξη, όπως πολύ σωστά είπαν οι προλαλήσαντες, μεταξύ άλλων ο κύριος Παρόσο. Έχουμε λοιπόν πολύ καλή απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Το ποιοι είναι οι καλύτεροι στόχοι δηλαδή για να δαπανίσουμε τα χρήματά μας. Το ε, σημαντικό αυτό στοιχείο είναι ακριβώς η πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντομπρόφσκι, πρόεδρος της Οικονομικής, Γεωργικής, Περιβαλλοντικής και Περιφερειακής Πολιτικής της Λετωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην ανακτήρια συνεδρία σήμερα το πρωί ε, εκπρόσωπος ε, του, της Προεδρίας ε, μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, και πάρα πολύ που άκουσα ότι η βασική αρχή είναι η ελεγγύη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, πολύ συχνά υπάρχει με μια απόκληση μεταξύ αρχών που εξαγγέλλονται και της πραγματικότητας. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ο προπολογισμό της Επιτροπής ε, περιλαμβάνει μια ε, περικοπή της τάξης του 600 αφορά το κονδύλια συνοχή στη χώρα μου. Μιλούμε για ε, περικοπές στα κονδύλια συνοχής σε μια από τις χώρες που δεν είναι μόνον φτωχή, αλλά έγινε ακόμα φτωχότερη τα τελευταία χρόνια. Ε, πώς μπορούμε να αποκαλέσουμε κάτι τέτοιο αλληλεγγύη. Πώς μπορώ εγώ να πάω στους ψηφοφόρους μου και να τους εξηγήσω αυτή τη μορφή αλληλεγγύη. Τι είδους αλληλεγγύη είναι αυτή. Και θα ήθελα να σας θέσω ευρύτερα το ερώτημα εδώ τι είδου Ευρώπη πρόκειται να οικοδομήσουμε. Θα οικοδομήσουμε μια Ευρώπη η οποία βασίζεται σε κάποιες κοινέ αξίες και αρχές ή θα οικοδομήσουμε μια Ευρώπη όπου ο καθένας κινείται ατομικά, όπου οι δυνατοί στραγγαλίζουν τους αδύναμους, τους φτωχού και τους μικρούς. Ε, βεβαίως η απάντηση της ερώτησης μοιάζει προφανής σε ένα ρητορικό επίπεδο. Αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την παλιά Σοφία. Ε, μπορείτε να εξαπατάτε ορισμένου ανθρώπους κάποτε, αλλά όχι τους, πάντο, τους πάντες συνεχώς. Θα πρέπει να ε, καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, γιατί η νομιμότητα της Ευρώπης στα μάτια των ψηφοφόρων συναρτάται από τη συνέπεια που επιδεικνύουμε σε σχέση με την προσήλωσή μας στις αρχές που έχουμε εξαγγείλει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντανούτα Χούμπνερ, ε, πρόεδρος της ε, Περιφερειακής ε, Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Θα θυμάστε ότι σήμερα το πρωί ο πρόεδρό μα, ο κύριο Μάρτιν Σούλτ, είπε ότι ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και Εθνικοί Προπολογισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται για να εκπληρώσουν του κοινού ευρωπαϊκού στόχου δημιουργία θέσεων απασχόληση με ένα συμπληρωματικό τρόπο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια αναπτύξαμε τη νέα οικονομική διακυβέρνηση, το σύστημα των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων για να συσφίξουμε του δεσμού μεταξύ Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και Εθνικών Προπολογισμών. Αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να δούμε το δυναμικό των πολιτικών που ε, περιέχονται ακριβώς στην ε, διασύνδεση αυτή μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων. Και πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός καταλήτης στην δημιουργία διαρθρωτικών αλλαγών και στην πυροδότηση της ανάπτυξης. Ε, σε συνάντηση με την πολιτική συνοχή. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω σχετίζεται με αυτή την αιμονή για, στην ε, έννοια της ανάπτυξης που έχουμε αναπτύξει τελευταία. Ε, κάθε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ισχυρίζεται ότι αυτό το πολιετές το δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει σαν βασικό στόχο την ανάπτυξη. Ωστόσο όλοι παρακολουθούμε τι ειδήσει από το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, διαβάσουμε τι εφημερίδες, διαβάσουμε τα πρακτικά των Ευρωπαϊκών Συνόδων, των Συνόδων κορυφή, και ξέρουμε ότι, όλοι, πολύ γνωστοί ευρωπαϊκοί ε, πολιτικοί ανταγωνίζονται ο ένας με τον άλλον όσον αφορά τις προτάσεις περί κοπών. Και όλα αυτά δεν συνάδουν με την ανάπτυξη. και ταυτόχρονα ισχυρίζονται ότι εξαγγέλουν κάποια υποστηρικτικά μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Επίσης λέγεται ότι είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή, η οποία έχει επιλεγεί και στοχευθεί για μακροοικονομικές ε, κυρώσεις. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα πρέπει να δούμε την πρόταση της Επιτροπής, η οποία προετοίμασε ένα πολύ καλά ισορροπημένο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, επικεντρωνόμενη στις ε, πολιτικές ανάπτυξης και επίσης έναν αξιοπρεπή προπολογισμό όσον αφορά την υποστήριξη των ε, μέτρων αύξησης των σόδων. Εάν λοιπόν οι περικοπές εφαρμόζονται ενάντια στις πολιτικές δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, θα χάσουμε αυτή την ισορροπία την οποία προτείνει η Επιτροπή και θα επιστρέψουμε στην ε, φιλοσοφία, στο σκεπτικό της δεκαετίας του 90 όσον αφορά τον προπολογισμό. Και ε, θεωρώ ότι είναι ένα μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πει όχι στις ε, περικοπές που σχετίζονται με τις δαπάνες για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χίμπνερ, η κυρία Ολοπέσκου, ε, από το Υπουργείο Εξωτερικών της ε, Ρουμανίας. Ευχαριστώ. Όλοι είπαμε ότι ο προπολογισμό πρέπει να είναι μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και την τόνωση τη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Επίση, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση τη κρίσης ε, του χρέους και να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Θεωρούμε ότι χωρίς επαρκή κονδύλια μετά το 2013 μόνο περιορισμένη συμβολή θα έχουμε στην εκπλήρωση και την επιδίωξη των ε, συμπεφωνημένων στόχων και της δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ λίγο θα σεβαστούμε την αρχή τη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία αναζητά μια δέσμη μέτρων που να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία. Διότι η πραγματικότητα τη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νέε ανάγκε ανάπτυξη στα κράτη-μέλη για να καλυφθούν τα κενά. Βάσει τη λιτότητα του προπολογισμού σήμερα, τα κονδύλια ανάπτυξη δεν μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αύξηση, την οικονομική αύξηση και τις επενδύσεις με επενδύσεις των κατώμελών από τα διευθυντικά ταμεία, από την αγροτική πολιτική. Πρέπει να ολοκληρώσουμε ακόμα την ενιαία αγορά. Η Ρουμανία είναι υπέρ της διατήρησης των σημερινών μορφών ευελιξίας που προβλέπονται στον προπολογισμό, που είναι βιώσιμη επίσης το ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι επιτρέπουν απαρκές πλαίσιο ελιγμών, μέσω του προπολογισμού και προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της νοσονομικής πειθαρχία και της κάλυψης των νέων αλλαγών που μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτα. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κροατίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μπρέγκοβιτς από το Κρατικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές της ημερίδας αυτής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που μας προσκάλεσαν σε αυτήν την συνάντηση ψηλού επίπεδου. Θέλω όλος ιδιαίτερος να ευχαριστήσω τον κύριο Σούλτ και τον κύριο Λαμασούρ για το θερμό του καλωσόρισμα χθε στο δείπνο που μας ε, παρέθεσαν. Σήμερα θα ήθελα ως βουλευτής από την Κροατία να μιλήσω και υπό την άλλη μου ιδιότητα ως μελλοντικού παρατηρητή από την Κροατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Κροατία πρόσφατα υπέγραψε τη συμφωνία ένταξής της και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως από την Ουγγαρία και την Πολωνία που μας βοήθησαν ιδιαίτερα. Θα ξέρετε ότι οργανώθηκε δημοψήφισμα στην Κροατία στις 22 Ιανουαρίου φέτος και τα δύο τρίτα της χώρα ψήφισε υπέρ τη ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διαδικασία αυτή χρειάστηκε να παρουσιάσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα στου πολίτες της χώρας. Δύσκολο ήταν να πετύχουμε στήριξη από τους πολίτες της Κροατίας για το ευρωπαϊκό εγχείρημα σε καιρού οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση και σε καιρού κρίση του ε, κατοικού χρέου. Κάτι που είδαμε να πλήττει πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε τα περασμένα χρόνια. Τώρα όμω, με τη σημερινή συζήτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή ευκαιρία. Όχι μόνο για να μελετήσουμε καλύτερα το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και για να δούμε πώ το πολιτικό σκηνικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βελτιωθεί χάρη στη συμβόλη του προπολογισμού. Πώ μπορούμε να διασυνδέσουμε τη λίστα προτεραιοτήτων του 2020 με ακριβώ το πολιτέ αυτό πλαίσιο πώς επίσης μπορούμε να συσχετίσουμε τις εθνικές ανάγκες με την κάλυψη των αναγκών του προπολογισμού. Να εξέλθουμε από την κρίση και να αναζητήσουμε μηχανισμούς αλληλεγγύης. Στην Κροατία δύο στοιχεία πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου για τη χώρα αυτή. Πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η συνθήκη ένταξης και κάτι άλλο που θα, θα χαρακτήριζα προσδοκίες, τις ε, φυσικές προσδοκίες, τις προσδοκίες που φυσικά προκύπτουν σε μια χώρα που πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια λοιπόν μέτρα λιτότητας σίγουρα χρειάζονται, όμως υπάρχουν και άλλες προσδοκίες. Ακόμη ε, θέλουμε οι πολιτικές συνοχής να διασυνδέονται με τις επενδύσεις, με την ε, ανάπτυξη και την έρευνα χαρτοφυλάκια κονδυλίων ε, σε ό,τι αφορά την γεωργία και άλλες επενδύσεις είναι στοιχεία που επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρίως για τη μεταβατική περίοδο. Ε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την προστασία των κοινών εξωτερικών συνόρων πλέον. Θα θέλαμε η φωνή μας να ακουστεί και σε αυτήν την περίπτωση και σε άλλα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι τώρα θα μιλάμε πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση με 28 μέλη. Σας ευχαριστούμε κυρία Λοκασέβιτσα, πρόεδρος της Επιτροπής από το Λετωνικό, ε, τη Λετωνική Γερουσία. Um, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που η Δανέζικη Προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε πέρσι το φθινόπωρο σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και που έχουν προσκληθεί και ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι εθνικέ κυβερνήσει. Συμφωνώ ε, απόλυτα με τις αρχές τις οποίες σκιαγράφησε η Δανή Πρωθυπουργό ε, στην ομιλία της. Ευχαριστώ πολύ ε, που παρέχεται το πλαίσιο για τη συζήτηση αυτή. Σύντομα να παρουσιάσω τη θέση της Λετωνίας ε, και του Κοινοβουλίου της για το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το επόμενο διάστημα προγραμματισμού και τις επιπτώσεις του για την ανταγωνιστικότητά μας. Η Λετωνία θέλει οικονομική ανάπτυξη. Είμαστε αυτή τη στιγμή χώρα που λαμβάνει πόρους, αλλά για να γίνουμε χώρα δότης ε, χρειαζόμαστε ε, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Γι' αυτό συμφωνούμε με ε, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, ωστόσο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποιες από τις λεπτομέρειες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, η πολιτική συνοχή η Λετωνία έχει εφαρμόσει τα σχετικά μέτρα με ε, υπεύθυνο τρόπο. Έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία και έχουμε εφαρμόσει τα μέτρα του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Πρωτού καλά, καλά γραφτεί αυτό και αυτό έχει ε, θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ μας τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε ότι Κατά την κατανομή των πόρων της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτά. Δυστυχώς όμως ε, βλέπουμε ότι το προτινόμενο ανώτατο όριο θα, σημαίνει, θα σημάνει ότι ε, κατά 20% θα μειωθούν οι πόροι συνοχής για την Λετωνία διότι ε, είχαμε ε, μείωση του ΑΕΠ ε, κατά 25% συσσωρευτικά. Ε, αυτό όμως δεν είναι υποστήριξη μιας χώρας που είναι υπέρ των ε, αυστηρών ε, δημοσιονομικών μέτρων. Ε, τα ταμεία συνοχής αποτελούν μέσο για την προσέλκυση επενδύσεων. Η οικονομική ανάπτυξη πέρσι ήταν 5,5%. Δεύτερον, ε, πολύ σύντομα για την κοινή γεωργική πολιτική. Δυστυχώς οι άμεσες ε, πληρωμές δεν ε, έχουν εισαχθεί βαθμία όπως είχε συμφωνηθεί κατά τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Λετωνοί Γεωργοί ακόμα συνεχίζουν να λαμβάνουν τις χαμηλότερες άμεσες πληρωμές ε, είναι τρεις-τέσσερις φορές χαμηλότερες από αυτές ε, των ε, ομολόγων τους σε άλλες χώρες. Αυτό αντίκειται στις κοινέ αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινή αγορά παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στους γεωργούς, μόνο όμως αν έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, η γνώση. Η γνώση αποτελεί σημαντική κινητήριο δύναμη της οικονομίας μας. Θα πρέπει να επιδιώκουμε ε, την αριστεία, θα πρέπει να στηρίζουμε την υποδομή για την επιστήμη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει τα κέντρα αριστείας να συγκεντρώνονται μόνο σε κάποιες χώρες. Ε, αυτό θα ήταν λάθος προσέγγιση. Ε, συνοψίζοντας, ε, η ισότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκοντας ε, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις αρχές αυτές όταν εκπονούμε το επόμενο, την επόμενη φάση του πολιετού σε δημοσιονομικού πλαισίου. Θα έχουμε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη αν μείνουμε στις αρχές αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώραν Φάρμ, Ευρωβουλευτής ε, της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι συντονιστής ε, των Σοσιαλδημοκρατών στο, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και εισηγητής των ομολόγων για τον project bonds, όπως ανέφερε ο, ο ε, Πρόεδρος στην εισαγωγή του. Ε, είμαι πολύ ευγνώμων προς την ε, Πρωθυπουργό Χέλε Τόνινγκ Σμιτ ε, για την ομιλία της σήμερα το πρωί, παρότι δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Καταρχήν μίλησε για τον εξυγχρονισμό του προϋπολογισμού με μετακίνηση προς την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Από ό,τι κατάλαβα όμως θα γίνονται από τις σχετικές περικοπές στην κυρία γεωργική πολιτική και τα διαφορετικά ταμεία. Ας επικεντρωθώ στα ταμεία συνοχής και τα διαφορετικά ταμεία. Ε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο τρόπο να πετύχουμε τον εξυγχρονισμό, να χρησιμοποιήσουμε τα διορθωτικά ταμεία ω μέσο για την καινοτομία, για τον εξυγχρονισμό, για την υποδομή και για τι επενδύσει. Ε, δεν υπάρχει άλλο μέσο το οποίο να είναι εξίσου αποτελεσματικό με τα διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά τι επενδύσει για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόληση σε μια χώρα που το χρειάζονται ω πράξη αλληλεγγύη που να επικεντρώνεται περισσότερο στι ε, λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ, λέει η Χερετόνιγκ Σμιτ και συμφωνώ με αυτό. Αυτό όμω ε, σημαίνει ότι τα ταμεία συνοχή θα διαγραφούν, θα καταρριθούν για, τις πιο πλούσια, για τα πιο πλούσια κρατημέλη. Δεν ε, είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει να γίνει αυτό και για αρκετού λόγου. Διότι και τα πιο πλούσια κρατημέλη έχουν μειονεκτικέ περιοχέ που χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην υποδομή, στην καινοτομία για την ε, ολοκλήρωση κλπ. Και χωρίς ε, την ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν νομίζω ότι θα λάβουν αποζημίωση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς αν χάσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση λόγω της οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αν καταργηθεί η χρηματοδότηση για τις ε, μειονεκτικές ε, περιοχές ε, πλούσιων χωρών, θα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει σε περιοχές όπως είναι η Ουαλία ή ο Βορράς της Σουηδίας, όπου ήδη το κλίμα είναι κάπως περίεργο. Τα διαρθρωτικά ταμεία επίσης παίζουν ρόλο για την διασυνοριακή και διεθνική συνεργασία. Ε, επίσης ε, θα ε, έχει κακές επιπτώσεις όσον αφορά την περιφερική τομή. Ε, ε, για, την, ε, για το Περιφερειακό Ταμείο. Η Χέρα Τόνι Σμιτ λέει επίση ότι θα πρέπει να κλείσουμε προγράμματα τα οποία δεν επιφέρουν αρκετή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εμεί είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε μια τέτοια συζήτηση παρότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι. Εάν όμω υπάρχουν κοινέ προτάσει του Συμβουλίου για το κλείσιμο προγραμμάτων είμαστε ανοιχτοί να γίνει μια τέτοια συζήτηση αλλά το πρόγραμμα μέχρι τώρα ήταν ότι δεν υπήρχαν τέτοιες προτάσεις από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν σχετικά με τι περικοπέ. και γι' αυτό προκαλώ τα κράτη-μέλη. Σας παρακαλώ, ε, παρουσιάστε μας αυτές τις προτάσεις για να τι συζητήσουμε σοβαρά. Η επόμενη ομιλήτρια είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Περιφερειών. I think we were told a few... Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είπαμε πριν από λίγα λεπτά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας στοιχίζει 67 απένες την μέρα, λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πω στους συναδέλφους εδώ ότι η γνωμοδότηση την οποία εγώ συνέταξα σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πέρασε από την Επιτροπή Περιφερειών τον Δεκέμβριο ομόφωνα με μόνο δύο ψήφους ε, κατά ε, από τον Βασίλειο. Κύριε White, θέστε το ερώτημα πόσο ε, τι φιλοδοξίε θα πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι στους Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερω φιλόδοξοι και θα πρέπει να στηρίξουμε τι προσδοκίε αυτέ στου προπολογισμού μα και θα πρέπει να του εφαρμόσουμε. Θα πρέπει να έχουμε ανάπτυξη ούτω ώστε να εξηγιάνουμε το δημόσιο χρέο ε, το οποίο έχει σωρευθεί τις ε, τελευταίες δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να το κάνουμε δεν, θα, δεν πρόκειται να επιτύχουμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει να έχουμε κάποια κίνητρα για τις ευιστάμενες επιχειρήσεις και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες επιχειρήσεις αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ε, τεράστιες συνεργασίες που δράσουν σε δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τράπεζες που έχουν δισεκατομμύρια ευρώ και δεν επενδύουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. πρόκειται να, από πού θα προέλθει αυτή η υποστήριξη, ε, η χρηματοδότηση. Κυρίες και κύριοι, εγώ πιστεύω ότι θα προέλθει από το Ταμείο Συνοχής και την χρηματοδότηση των διευθυντικών ταμείων, γιατί μόνο έτσι μπορούν να δοθούν κίνητρα στην ανάπτυξη. Και τώρα μπορώ να δώσω μια απάντηση στην ερώτηση κυρία Σέιμ, η οποία είπε τι πετυχαίνει αυτός ο προπολογισμό. Και θα ήθελα να σας το πω ε, ε, σε σχέση με μια περιφέρεια που έχει ένα πληθυσμό του 2,1 εκατομμύρια. Ε, από το 2000 τα επίσημα νούμερα δείχνουν ότι η πολιτική συνοχή και τα διορθωτικά ταμεία δημιούργησαν ένα πλεόνασμα 90.000 θέσεων εργασία και ένα πλεόνασμα 7.000 επιχειρήσεων και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, καταρτίστηκαν και ε, δημιουργήθηκαν 26.000 ευκαιρίες για επιχειρήσεις προκειμένου να επεκταθούν. Ε, και αυτό σε μια επιχείρηση, ε, σε μια περιοχή, συγγνώμη, 1,2 ε, εκατομμυρίων. Και έγιναν και μπορώντας να με τη δυνατότητα να δαπανίσουν οι άνθρωποι αυτοί αγόρασαν ε, ολλανδικά αγροτικά προϊόντα, Φιλανδέζικα κινητά και Ολλανδικά έπιπλα, καθώς και Ιταλικά ρούχα και πάρα πολλά άλλα πράγματα, κάτι που βοηθάει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Ο κύριος Μπαρόζο είπε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινωνία, ε, κοινότητα. Εμείς, ε, θα έλεγα, είμαστε μια Ευρώπη κοινοτήτων και μπορούμε να ευεργετηθούμε μόνο από την πολιτική συνοχή και μόνο εφόσον το κάνουμε θα στεφθούν οι προσπάθειές μας με επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ να ε, παραμείνετε στο χρόνο σας, να τηρήσετε τα χρονικά σα περιθώρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ την παρέμβασή μου παίρνοντα αφορμή από την παρατήρηση του κυρίου White, όταν είπε ότι ο προπολογισμό πρέπει να είναι ένας επενδυτικός προπολογισμός. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επικεντρώνεται στις δαπάνες και τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις οικονομίες μας, να τις κάνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε μια περίοδο κρίσης και εκεί χρειαζόμαστε μια κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη. Ένα καλό ε, πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να μας το δώσει η πολιτική συνοχής ως λύση. Εάν η πολιτική συνοχής ε, γίνει μια πολιτική για το μέλλον, Νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά ε, στο ερώτημα εάν θα έχουμε ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ναι, μπορούμε να έχουμε, μπορούμε να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη και κοινωνικά και εδαφικά. Όμω θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που τα θεωρώ κρίσιμη σημασία μεταξύ των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, τα κονδύλια για την ε, συνοχή. Το να μειωθούν το 40 δις το μηχανισμό για να Ε, να πρικοδοτήσουμε το πρόγραμμα Connecting Europe σημαίνει ότι θα κατέβουμε από 348 μέχρι στα 336. Όμως, τα κονδύλια των διαδοτικών ταμείων θα πρέπει να επιτρέψουν την εξισορρόπηση δημοσίων και ιδιωτικών ε, κονδυλίων που σε πολλές περιοχές της Ευρώπης επιτρέπουν ε, να υπάρξουν δημιουργήσεις θέσεις απασχόλησης και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης για τις ενδιάμεσες περιφέρειες που δημιουργούνται ως κατηγορία. Σε κάποιες ευημερούσες χώρες ε, υπάρχει στρέβλωση της ε, χρήσης της πολιτικής συνοχής σαν να ήταν αναδιαναμητική. Η αποστολή που έχει αναλάβει. Εδώ πρέπει να δούμε ξανά τις συνθήκες, διότι η ανάπτυξη σε περιοχές καθυστερημένες ως προς την ε, οικονομική αύξηση θα πρέπει και την ευημερία των πολιτών συνολικά να δούμε ότι ωφελούν και βεβαίως μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βιωτικά προβλήματα. Άλλο κρίσιμο σημείο είναι το λεγόμενο κάπινγκ. Εδώ θα διαφωνήσω με τον Ούγκρο ε, Υπουργό εδώ. Μιλάμε για ένα όριο 2,5% του ΑΕΠ. Για να παραμείνει ζωντανός ο επαρχιακός χαρακτήρας των πολιτικών ε, συνοχής θα πρέπει αυτό το όριο να μειωθεί ώστε να υπάρχει ισοδυναμότερη κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των ε, περιφερειών που χρειάζονται ανάπτυξη. Τις ερχόμενες ημέρες θα εγκρίνει έγγραφο ε, με, την, με τον ίδιο ε, το Ιταλικό Κοινοβούλιο που θα ζητούμε για το δημοσιονομικό πολιτές πλαίσιο ανακατανομή. Ευχαριστούμε κύριο Χουμπαρτσόν από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Eh, θα πω μερικά πράγματα πολύ σύντομα σχετικά με την θέση της Σουηδία ε, και του Σουηδικού Κοινοβουλίου όσον αφορά το ε, μακροπρόθεσμο προπολογισμό. Ε, θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι ε, τα κόμματα στο Κοινοβούλιο της Σουηδίας συμφωνούν όσον αφορά τις βασικές γραμμές, παρότι υπάρχουν φυσικά διαφορές όταν μπούμε στις λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε να περικόψουμε τον προϋπολογισμό. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι σημαντικό να έχουμε ε, ισχυρή πολιτική συνοχής. Έχουμε όμως ε, κάπως πιο περιοριστική ε, θέση όσον αφορά την ανάπτυξη του προϋπολογισμού. Θέλουμε δηλαδή πάνω από όλα εξυγχρονισμό του προϋπολογισμού. Και όπως είπαν ουσιαστικά και όλοι οι άλλοι ομιλητές στην αίθουσα τούτη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, ε, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ε, στις διασυνοριακές δομές. Αυτή η εξέλιξη όμως θα πρέπει να γίνει με εξυγχρονισμό, με αλλαγή των προαιροτήτων και εξοικονόμηση σε άλλους τομείς και με πιο καλή αποτελεσματικότητα θα σχολιάσω κάποια από τα επιχειρήματα κατά της θέσης μας. Ε, ένα είναι ότι δεν έχει ε, αναπτυχθεί, δεν, είχε δεν είδαμε τις ίδιες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όπως είδαμε με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ε, αλλά η Ευρώπη πρέπει να στέκεται στα πόδια της και πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό που να στέκεται στα πόδια του οι εθνικοί ε, προϋπολογισμοί πρέπει να καλύπτουν θέματα όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση ε, κλπ. Και μάλιστα ε, τα κράτη-μέλη έχουν την βασική ευθύνη για την πολιτική ανάπτυξης και απασχόλησης. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει από, τον, από, την οικονομική κρίση με την ε, μονομερή πολιτική λιτότητα που βλέπουμε. Ε, άσχετα από το τι ε, γίνει με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι ένα άλλο επιχείρημα για ε, αυξημένο προϋπολογισμό. Ε, ένα πολύ καλό επιχείρημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα αυξημένα καθήκοντα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το, όταν ε, αποκτά κανείς νέα καθήκοντα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να πληρεί και τα παλιά. Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα εξυγχρονισμό του προϋπολογισμού και πιο αποτελεσματική χρήση το Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σεβερά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι αυτή η ε, συγκέντρωση θα μας οδηγήσει στο συμπεράσμα ότι η ανάπτυξη είναι και ευρωπαϊκή φιλοδοξία αλλά και εθνική. Η ασφάλεια στην ευρύτερη της έννοια που συμπεριλαμβάνει και την κοινωνική και την οικονομική ασφάλεια είναι κάτι το αδιέρετο. Θα πρέπει λοιπόν το καθένα κράτος μέλος ξεχωριστά, το καθένα εθνικό κράτος μέλος να ενδιαφερθεί για τις οικονομικές, ε, την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Διότι οι διαχωρισμοί ε, αυτού του τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν ένα αμφιβόλο και ε, πλήττουν την ακαιρεότητα ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του καθενό κράτου μέλου ξεχωριστά. Θέλω εδώ να τονίσω ότι ο προπολογισμό τη πολιτική συνοχή διαρκώ είναι αντικείμενο επιθέσεων. Επιθέσεων που υποκρύπτουν τους παλιούς δαίμονες αντιπαλωτήτων μεταξύ των κρατών και λαϊκιστικών προσεγγίσεων. Η τάση να μειωθούν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής είναι ένα από τα πιο φρικτά παραδείγματα αυτής της πραγματικότητας. Υπάρχει και η άποψη ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η θέση προτεραιοτήτων και η αιρεσιμότητα στην ε, απόδοση των κονδυλίων. Όμως οι μακροοικονομικές συνθήκες καθώς ε, και οι επιδόσεις θα έπρεπε να διέπουν το πνεύμα της πολιτικής ε, συνοχής και τα κριτήρια της. Τα κράτη που περισσότερο χρειάζονται κονδύλια συνοχής είναι ακριβώς εκείνα που έχουν προβληματικές μακροοικονομικές επιδόσεις. Επίσης έχουν τις περισσότερες δυσκολίες στο να δώσουν καλά αποτελέσματα, καλά προγράμματα. Άρα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι εμείς θα πρέπει να κινητοποιήσουμε μηχανισμούς που πραγματικά θα βοηθήσουν τα κράτη που χρειάζονται κονδύλια και όχι να τα κατευθύνουμε σε όσους είναι ήδη ανεπτυγμένοι, οπότε έχουν και ευκολότερη πρόσβαση στα καμπύλια. Η διευκόλυνση για τη διασύνδεση τη Ευρώπη είναι ένα καλό παράδειγμα, μια καλή ιδέα μεταξύ των όσων ελέγχθησαν και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χρηματοδοτεί τον εαυτό μέσο με 40 δι ευρώ συν 10, τα οποία θα πάρει από το Ταμείο Συνοχή. Όμω, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αναλογικά θα έχουν βάσει του Ταμείου Συνοχή οι χώρε με το υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότηση ακριβώ και τη μεγαλύτερη στήριξη για αυτό το νέο πακέτο μέτρων. Χρειαζόμαστε λοιπόν διασφαλίσεις ότι τα εθνικά χαρτοφυλάκια θα ε, ανταποκρίνονται ε, στις ανάγκες της υλοποίησης και να αποφύγουμε να υπάρξουν εντυμένοι. Δηλαδή, οι χώρες που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη από το Ταμείο Συνοχής. Ακριβώς αυτές δεν έχουν τις απαραίτητες διοικητικές δυνατότητες. Τελευταίο παράδειγμα, το να παραμείνουν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής στο 2,5% του ΑΕΠ ασχέτως με το επίπεδο ανάπτυξης ε, στα κάτι μέλη και αυτό είναι παράλογο. Η ιδέα αυτή ουσιαστικά είναι μια πραγματική ριζοσπαστική μείωση και με αυτή την πρόταση κλείνω μια ριζοσπαστική μείωση που αγνοεί την αρχή της αλληλεγγύης και η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής συνοχής. Κάτι που ε, είναι αδύνατο σε μια χώρα, μπορεί σε μια άλλη να ισχύει. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό, είπε ο Κέιν. Ευχαριστώ. Από την Κροατική Βουλή, ο κ. Ζουρκοβίτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ιδανική Προεδρία αξίζουν συγχαρητήρια για να θέσουν προποθέσει μια επιτυχία. Η Κροατία ε, έχει διδαχθεί τι σημαίνει κρίση με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο. Και, αλλά μάθαμε ότι κατά τη διάρκεια, ε, ότι μια τέτοιου είδου κρίση μπορεί να ξεπεραστεί. Πώ μπορούμε τώρα να οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον με την αύξηση του διαλόγου, με ενότητα, αλληλεγγύη και εξισορρόπηση των ε, δαπανών. Η Κροατία συμμερίζεται τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει ευνοϊκέ προποθέσει για την ανάπτυξη επενδύσεων και την απασχόληση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πρόταση τη Επιτροπή για ένα νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι εξισορροπημένη και ρεαλιστική. Ιδιαίτερα όσον αφορά τι συζητήσει που επικεντρώνονται στην πολιτική συνοχή, στην πολιτική και την πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η σταθερότητα χρειάζεται στεναρή υποστήριξη. Ε, ελπίζουμε ότι όλες οι δυνάμεις θα συσπηρωθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σιδωνία, Σιδωνία Γιαβαλέσκα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συνάδελφοί μου από την Επιτροπή Προπολογισμών με ενθάρρυνε να μιλήσω γαλλικά, αλλά δεν είμαι έτοιμη να το κάνω. Ε, θα μιλήσω λοιπόν στα πολωνικά. Ναι. Εάν ε, θέλουμε να διατηρήσουμε τον παρόντα προπολογισμό και την ε, υφιστάμενη, δομή του, θα πρέπει να πω ότι ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές προσέγγισαν αυτό το θέμα. Δόθηκαν κάποια επιχειρήματα για το γεγονός ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να κατατείνει στην ανάπτυξη, τη μεγέθυνση. Θα ήθελα να υποφελθώ εδώ από την παρουσία σας και να κάνω μια έκκληση προς τους συναδέλφους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων προκειμένου να συνεργαστούν ούτω ώστε να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη χώρα μου, ενώ των ψηφόρων μου, συνειδητοποιώ ότι το ζήτημα δεν είναι πόσο δεν είναι τόσο η ποσότητα των κονδυλίων που είναι διαθέσιμα, αλλά περισσότερο ποιες είναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι μηχανισμοί μέσα των οποίων διοχετεύονται αυτά τα χρήματα. Και νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να μετακυλήσουμε το διοικητικό άχθος από τους ε, δικαιούχους ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια τα οποία δικαιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει αναφερθεί αλλά θεωρώ ότι αξίζει της προσοχής μας είναι το εξή. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες πτυχές του προϋπολογισμού. Θα πρέπει ε, να δούμε και ποια είναι τα άλλα κονδύλια, όχι μόνο αυτά από το Ταμείο Συνοχής, αλλά για παράδειγμα τι γίνεται με την εκπαίδευση, με την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτά είναι μικρότερα κονδύλια, αλλά άμεσα ή έμεσα τα κονδύλια αυτά ε, είναι εξαιρετικά χρήσιμα γιατί ενισχύουν τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων προκειμένου να έλθουν στην ε, αγορά εργασίας. Επίσης συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας, διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και νομίζω και θα πρέπει να διευκρινίσουμε και το ρόλο αυτής της μορφής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Και εάν δούμε τον αριθμό των δικαιούχων, διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετά περιορισμένος. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στην κινητικότητα. Και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους μικρότερους προϋπολογισμούς. Η κυρία Ελένα Αντρέ από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν. Ήθελα και εγώ να σχολιάσω τα θέματα που μας απασχολούν διότι η κατάσταση της Ευρώπης σήμερα δεν είναι απλή. Η κρίση του ευρώ έχει κάπως αντιμετωπιστεί, είναι σταθερή κατάσταση αλλά δεν έχει επιληθεί. Οι περικοπές στους εθνικούς προλογισμού είναι σοβαρές, τα μέτρα λιτότητας έχουν ε, σοβαρές συνέπειες στην οικονομία, την απασχόληση και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών αλλά υπάρχει και ένας παράγοντας τον οποίο ένα, διαφορές, μια διαφορά τον θίξαμε και εδώ στην αίθουσα την ανάκτηση της εμπιστοσύνη των πολιτών δεν στηρίζουν όπως προηγουμένως το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ακριβώς ε, για τους προηγούμενους παράγοντες που ανέφερα θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι δυνατότητα έχουμε με ρωμαλαία αντιμετώπιση να αντιμετωπίσουμε την κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι που ως τώρα δεν έχει γίνει επαρκώς. Και θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε στα θεμέλια μάλιστα της οικοδόμησης του ευρωπαϊκού ε, εγχείρηματο. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό μπορεί να μας βοηθήσει ως εργαλείο να ε, ενισχύσουμε την απασχόληση, την ανάπτυξη και να ξαναδούμε τις εθνικές δημοσιονομικές ε, προτάσεις. Αυτά που μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αφορούν κυρίως τις πολιτικές που στηρίζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως ακριβώς ο προπολογισμό μπορεί να προωθήσει και την ε, ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια και την κινητικότητα στην Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Ελπίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεχίσει να τηρεί υπηκοδομητική ε, θέση και να παρεμβαίνει ενεργά στη, συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα του προπολογισμού. Ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ή άλλως, είναι αρκετά συγκατημένος ώστε να θεωρηθεί οικονομικά ε, επαχθή. Άρα, γι' αυτό, Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την άποψή μου οι διαπραγματεύσει δεν μπορεί να επικεντρώνονται στη διατήρηση τη υπάρχουσα κατάσταση και στι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι φιλοδοξίε μα. Δεν μπορεί να στοχεύουν τα, τα συμφέροντα μόνο των πολυεθνικών. Διότι υπάρχει πρόβλημα με την αιμορραγία των φορολογουμένων. Θα πρέπει να υπάρξει επανεθνικοποίηση των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών, μεταξύ των οποίων η πολιτική συνοχής και οι υπόλοιπε πολιτικές του δημοσιονομικού πλαισίου. Γι' αυτό θα πρέπει να τονώσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και για το παρόν και για το μέλλον. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ε, και συνοχή ανταγωνιστικότητα. Και θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα τέτοιο ε, παγκόσμιο σκηνικό. Ο κύριος Όρμελ από τις κατοχώρες. Ως μέλος ε, του Ολλανδικού Κοινοβουλίου σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, η Ολλανδία ε, είναι αφησιωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε η Ευρώπη να περάσει τις διεθνείς προκλήσεις. Η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει. Ε, και άλλωστε βλέπουμε εδώ πέρα μια ε, Ευρωπαία νικήτρια στο πρόσωπο της κυρίας Κρούς που βρίσκεται εδώ. Ωστόσο βρισκόμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τρόπο νυφάλιο. Αποτελεί πρόκληση να ε, ανακαλύψουμε τι θα είναι καλύτερο να κάνουμε μαζί στην Ευρώπη, τι θα πρέπει να κάνουν τα κυρίαρχα κράτη-μέλη και τι οι τοπικές κοινότητες, επικουρικότητα με άλλα λόγια. Ε, όσον αφορά την γραφειοκρατία θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Οι κάτω χώρε ε, καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρει λύση ε, σχετικά με το μηνιαίο τσίρκο, το ταξίδι ε, στο Στρασβούργο. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό στους ψηφοφόρου μου και είναι αρνητικό για την ευρωπαϊκή εικόνα. Καλούμε την Κομισιόν να περικόψει τον προϋπολογισμό της διοίκησης αντί να τον αυξάνει. Αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Έχουμε την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, την Frontex, ε, την Κοινοτομία, τη Γεωργία, την Πολιτική Ενέργεια, στο, την αλλαγή του κλίματο. Φυσικά απαιτούνται χρήματα για όλα αυτά. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα για να αυξήσει τη συνέργεια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του εθνικού προπολογισμού. Να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Ε, με ένα σπάρο δύο τριγώνια ακούτε ότι ε, <laughs> δεν είμαι ε, μέλος του κόμματος των φιλόζων στο κοινοβούλιο μου είναι πιο εύκολο να επενδύουμε όταν βλέπουμε τις εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο, ε, επενδύοντας στις κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια και ο έλεγχος είναι απολύτως απαραίτητα για την νομιμότητα των δαπανών μας. Δεν έχουμε ακόμα λάβει τις ε, εθνικές εκθέσεις ε, δαπανών από όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνέργεια, αλληλεγγύη, ε, ε, συνέργεια, αλληλεγγύη επικουρικότητα για να πάει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομίας της Ισπανίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τίθεν να όσον αφορά την ευρωπαϊκή ελοκλήρωση και βεβαίω το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπει όλες τις προσπάθειες θα πρέπει να υπάρξει ένα σωστός, ε, ε, σωστός προσανατολισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τις ε, δαπάνες που γίνονται εξ ονόματος της αλληλεγγύης και της όφησης προς την ανάκαμψη και την της ευημερίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, υπό την έννοια αυτή μα ενισχύουν πάρα πολύ τρει πολιτικές. Πρωτίστως η κοινή αγροτική πολιτική, την οποία υπερασπιζόμαστε στεναρά. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι μια ισχυρή πολιτική, να έχει επαρκείς ε, πόρους. Επίσης, όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, ε, θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη αναγνώριση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της ε, γεωργικής ε, πολιτικής. Δηλαδή θα πρέπει να ενισχύει επίση την εσωτερική αγορά και να διασφαλίζει, εξασφαλίζει την ψηφιστική ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων και να υπάρξει μια προσπάθεια αντιστροφή τη κλιματικής αλλαγής. Είναι σίγουρο ότι ορισμένε πρόσφατες εξελίξει έχουν σημαντικέ επιπτώσει στην κοινή γνώμη τη Ισπανίας και μα οδηγούν να υποστηρίξουμε στεναρά τη δημιουργία ενό αποθυματικού για τι γεωργικέ κρίσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να παρακαμφθεί στι μελλοντικέ συζητήσει σε σχέση με τον προπολογισμό. Κατά δεύτερο λόγο, η Ισπανία, η οποία αναμφίβολο ήταν, ε, επωφελήθηκε πάρα πολύ από την πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό τη επέτρεψε να συσσωρεύσει ε, ε, να ενισχύσει μάλλον τις υποδομές της και να οδηγηθεί στη σημερινή τη ευημερία επιθυμεί την ε, συνέχιση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ε, εξελίσσεται αυτή η πολιτική συνοχή και αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια εκ νέου επικαιροποίηση των στόχων της και θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαχείριση των κονδυλίων και να υπάρχει μια σωστή χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε τις ενδιάμεσες ε, περιφέρειες οι οποίες ε, ε, δεν εμπίπτουν στις ζώνες σύγκλησης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται, να εξελιχθούν προς τις πιο εξελιγμένες ζώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τρίτο λόγο, θα ήθελα να δώσω έμφαση στις πολιτικές που προσανατολίζονται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς που, μας, ε, που να μας επιτρέπουν να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την ευημερία σε όλες τις χώρες. Η αριστεία θα πρέπει να είναι ένας ε, σκοπός αυτός καθ' αυτό. Ε, και θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε μια κλίμακα προς την αριστερία, ούτως ώστε, ούτως ώστε όλες ε, οι χώρες μέλη να μπορούν να ε, να μπορεί να του προσφυγή σε αυτά τα κονδύλια που προορίζονται για την αριστεία. Θα πρέπει επίση να ενισχύουν οι μικρομεσαίε υποχειρήσεις από την έννοια αυτή. Ε, πιστεύω ότι η σύγκληση τέτοιου είδου συνεδρίες που επιτρέπει μια προσέγγιση των Εθνικών Κοινοβουλίων στι συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην, ε, Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερω χρήσιμε όσον αφορά και μια μελλοντική προσέγγιση των διαφόρων ε, θεωρήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. από, την, από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα ελέγχθησαν και σκέφτηκα με ποιο μήνυμα θα επιστρέψει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή τη δεύτερη ε, διοργάνωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, ούτε ώστε να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτή την κρίση και να εξασφαλίσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε η σύντηση περί λιτότητας να γίνεται μόνο σε εθνικό επίπεδο και η πολιτική δαπανών και ανάπτυξης να γίνεται αποκλειστικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να σκεφτούμε από κοινού πού θέλουμε να επενδύσουμε, σε ποιου τομεί ακριβώ θέλουμε να γίνουν οι επενδύσει. Μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντοτε μια επενδυτική πολιτική. Αλλά θα πρέπει επίση να θέσει κάποιε προτεραιότητε. Πολλέ προτεραιότητε είναι αναγνωρίσιμε. Για παράδειγμα, στην ε, Αυστρία συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε κάποιες διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, αλλά μελλοντικά θέλουμε να επενδύσουμε στην ε, εκπαίδευση, στην ε, ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία. Και αυτό μπορούμε να το ξαναδούμε να αντανακλάται μέρη και στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο περίγραμμα, δηλαδή ε, πού θα συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξοικονόμηση και σε ποιους ε, τομεί θα πει ότι χρειαζόμαστε αυτές τις επενδύσεις για την εκπαίδευση, για την επιστήμη, για την καινοτομία, για ε, σε σχέση με το μέλλον. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσει ο προπολογισμό έτσι που ε, θέματα τα οποία ε, αφορούν πολλά κεφάλαια του προϋπολογισμού να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα για να δούμε πού θέλουμε ακριβώς να δώσουμε όθηση για αυτούς τους ε, τομείς. Η κυρία Κρούς αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε ε, έχοντας κατά νου συγκεκριμένε ε, διοικητικές ε, μεταρρυθμίσεις, μείωση της γραφειοκρατίας κλπ, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι να επιβεβαστούμε στο ίδιο πλοίο εν σχέση με την, τον προσεκπλήρωση στόχο της εξασφάλισης των μελλοντικών γενεών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντουάρτε Πασέκο από την Πορτογαλική Βουλή. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας ότι αν από όλα αυτά που λέμε κάτι μπορούμε να συμπεράνουμε, ιδίω μας ακούσαμε να λένε οι ευρωβουλευτές, είναι ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση. Μέσα από όλες τις παρεμβάσεις, τουλάχιστον σε δύο σημεία. Από τη μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτέ θα πρέπει να είναι οι πρώτε οι στρατηγικέ για να διατρανώσουμε τι αρχέ που περιλαμβάνει και η συνθήκη, δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ακριβώ τη στρατηγική αυτή για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης θα πρέπει να έχει κατάλληλες ε, διαστάσεις και προπολογισμό. Ιδάλλως θα έχουμε μια παράλληλη αντίφαση. Και θα πρέπει η ανάπτυξη αυτή η αύξηση του προπολογισμού να γίνει μέσω αλληλεγγύης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πρέπει να δούμε ότι η συνοχή λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Και το ίδιο και οι επενδύσεις που προκύπτουν από τη συνοχή, προκειμένου να πετύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο. Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό διότι υπάρχει και η άποψη ότι οι επενδύσεις που γίνονται μέσω της πολιτικής συνοχής δεν είναι επενδύσεις που θα πρέπει να ωφελούν μερικούς μόνον. Όχι. Η άποψη που πρέπει να υπερισχύσει είναι ότι ωφελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Διότι υπάρχουν ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν πραγματικά δυνατότητε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνέ επίπεδο. Μόνο η ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να κερδίσει. Και οι επενδύσεις στις υποδομές, στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, είναι προφανώς επενδύσεις που έρχονται να τονώσουν ακριβώ την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, Πρόεδρε, και εμείς ε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε η, το, ανάπτυξη και η συνοχή να γίνουν οι δύο όψει του ίδιου νομίσματο. Αυτό θέλουμε να περασπιστούμε πάνω από όλα εδώ. Κυρία Σέντερ, Ευρωβουλευτή για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ που έγινε αυτή η συνεδρίαση ως συνηγήτρια της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Ε, χαίρομαι που μπορούμε στο πλαίσιο της συνάντησης να ακούσουμε τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, υπό την έννοια αυτή, ε, υπό την έννοια του εξευρωπαϊσμού των ε, εσόδων και να προσδώσουμε μια ευρωπαϊκή πτυχή όσον αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ε, σε σχέση με το άρθρο 311 που συνδέεται με την ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων και των υπηρεσιών διατυπώνεται μια ε, πολύ σημαντική εντολή από την οποία ευεργετούνται όχι μόνο οι χώρες μέλη αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών δεν έχουν ε, επενδύσει αρκετά σε αυτή την έννοια της κινητικότητας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί εθνικοί εγωισμοί που παρεμποδίζουν την κινητικότητα. Και ε, θα ήθελα να σε επενθυμίσω το τελευταίο ε, δράμα το οποίο ζήσαμε στις δημοσιονομικές πρακτικές 2012 και 2013. Και όπως είπε η κυρία Κρούσε, υπάρχει μία ε, είδαμε τι έγινε με την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία που οι στάχτες της έκρηξης παρέλυσαν τις συγκοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πρόταση για την Connecting Europe Facility η οποία έρχεται με 20 χρόνια καθυστέρηση, γιατί ήδη η Λευκή Βίβλος ε, έδινε έμφαση σε μια ανάπτυξη κινητικότητας μέσω βελτίωσης των υποδομών. Ε, αυτή τη στιγμή της ε, κρίσης υπάρχουν άλλες περιοχές όπως είναι η Βραζιλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα που επενδύουν ε, στις υποδομές ούτως ώστε να αυξήσουν την κινητικότητα. Το Connecting Europe ε, Facility είναι ένα στίχημα για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και νομίζω ότι θα ε, συμβάλλει στην αύξηση της ευρωπαϊκής συνοχής και στο ξεπέρασμα των εμποδίων που παρακολύουν το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Επίσης θέλουμε να συνδέσουμε και ε, τις, τους αερολιμένες. Ε, ζητούμε επιπτώσει συνέργειας μεταξύ των συγκοινωνιών και θέλουμε να βελτιώσουμε και την ε, αστική κινητικότητα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, ούτε ώστε να ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα. Και όλα αυτά για να δώσουμε μία όθηση στην ευρωπαϊκή ανάκαμψη και να αποδεσμεύσουμε πολλές μεμονωμένες περιοχές που δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την απασχόληση. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ανάγκη της, του εξυγχρονισμού των υποδομών της κινητικότητας με έναν βιώσιμο και ποιοτικό τρόπο, ούτε ώστε να ξεπεραστούν τα σύνορα και να ελοπίσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν επιτρέπεται να παραλύει από την έκρηξη ενός ηφαιστείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ορθανοκράτη από το ε, Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι συμμετέχοντες, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, στο σημερινό φόρουμ. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με την ε, πολιτική συνοχή. χωρί να χρειαστεί να επαναλάβω όσα είπαν οι προλαλήσαντε. Καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω για την κοινωνική συνοχή. Ε, η επιχειρηματολογία μου στηρίζεται στις ε, σκέψεις ε, του κυρίου White. Ε, σήμερα το πρωί τέθηκε επανειλημμένα το ερώτημα εάν μπορεί να περιμένει κανείς από τον Ευρωπαίο πολίτη να πληρώνει περισσότερα χρήματα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να περιμένουμε από τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ε, ε, συνέπειες της κρίσης να πληρώνουν περισσότερα. Ε, δεν είναι πια τόσο ενθουσιασμένοι με την Ευρώπη οι πολίτες αυτοί. Ήδη έχουν κάνει θυσίες για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Βλέπουν όμως ότι άλλοι κερδίσανε ενώ οι ίδιοι έχασαν. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε η πολιτική συνοχής Ε, και οι πόροι της να μειωθούν και να αφήσουμε ξεκρέμαστους αυτούς που υποφέρουν περισσότερο. Όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ισούται με τον προϋπολογισμό της, τότε οι πολίτες αυτοί θα σκεφτούν ότι αν ε, γίνουν περικοπέ ε, στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα σκεφτούν ότι θα λάβουν ακόμα λιγότερα και ε, όταν ο κόσμος απογοητεύεται βλέπουμε ενίσχυση των ακροδεξιών δυνάμεων και τότε θα βρεθεί σε κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα θα είναι πολύ σημαντικότερη κρίση εάν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ακροδεξιές ε, οργανώσεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να ε, διατηρήσουμε την υποστήριξη των πολιτών από το να πρέπει να ε, τους ξανακερδίσουμε μετά την ανάδειξη της ακροδεξιάς. Ο μικρότερος προϋπολογισμός οδηγεί σε μείωση της εμπιστοσύνης και μείωση της αλληλεγγύης. Ουσιαστικά δηλαδή μείωση της διάθεσης για συνεργασία θεωρούμε απαράδεκτο να μειώσουμε κατά 20% τους, ε, τα ταμεία. Η Ουγγαρία παραμένει ε, σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πιστεύουμε όμως ότι η κυρία Ντανούτα Χιούπνερ έχει δίκιο όταν υπερασπίζεται την πολιτική αυτή. Η κυρία Χέρτσοκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η ιδέα που οργανώσαμε τη διάσκεψη αυτή. Μιλώ ως η συγγήτρια της Επιτροπής για Βιομηχανίας. Να ξεκινήσω από την αγαπημένη μου φράση. Τίποτα δεν μας ε, δίνει περισσότερες ελπίδες ε, στη ζωή μας από τις πρώτες 24 ώρες ε, μιας δίαιτας. Μετά το πρώτο 24ωρο όμως ανακαλύπτει κανείς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει κανείς απλά μη τρώγοντας, θα πρέπει να αθλείται κιόλα. το, τελευταίο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσαμε για τη δίαιτα, τη λιτότητα. πρέπει όμως να αθλούμαστε κιόλα. Αυτό σημαίνει τρεις βασικοί τομείς στον τομέα της βιομηχανίας. Καταρχήν, ο τομέας ε, ενέργειας ε, και τεχνολογιών ε, επικοινωνίας και πληροφορική. Όχι όμως τον χθεσινό τομέα, τον τομέα αυτόν για το μέλλον. Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες για να είμαστε διασυνδεδεμένοι και γι' αυτό χρειαζόμαστε το δεύτερο άθλημα, έρευνα, ανάπτυξη και, και καινοτομία. Με άλλα λόγια, ορίζον 2020. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν τα μέρη να ε, υποστηρίξουν αυτά τα αθλήματα. Είχαμε σχετική ε, διάσκεψη αυτή την εβδομάδα και υπόθηκε σαφώς ότι η επιστημονική αριστεία μαζί με την αριστεία στον τομέα της τεχνολογίας θα αποτελέσουν βάση οικονομικής αριστείας για το μέλλον και θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό όταν αθλούμαστε. Χρειαζόμαστε πολιτική διαστήματος, χρειαζόμαστε τον Γαλιλαίο, το GMS ε, και νέες τεχνολογίες τρίτο άθλημα που χρειαζόμαστε είναι βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει καταρχήν παραγωγή εντός της Ευρώπης, διότι το δεύτερο κύμα ε, καινοτομίας ε, και τεχνονοσία θα έρθει από ε, τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα ταμεία γι' αυτό. Και επίσης μιλάμε για τη νέα πολιτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νέα και τα παλιά κράτη-μέλη παντού. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτού που λένε ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη, χρειαζόμαστε όμως μια Ευρώπη για όλους. Εμείς οι Ευρωπαίοι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές διαφωνούμε ότι οι μακροοικονομικές προκλήσεις ε, μπορούν να καταπολεμηθούν με αφαίρεση πόρων από ε, τις ε, πολιτικές συνοχές. Θέλουμε να έχουμε ψηφιακή Ευρώπη για όλους, σε μια Ευρώπη για όλους θέλουμε να έχουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάρις Βόλσκι, μέλος του Κοινοβουλίου από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ζητήματα θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα το μέγεθος του προπολογισμού. Είναι μικρό, δεν αρκεί, αλλά υπάρχει και άλλος παράλληλος προπολογισμός, πολύ γενναιόδωρος συγκριτικά. Και εδώ έχουμε δύο επίπεδα αλληλεγγύης. Ένα της Ευρώπης των 27, 1% του ευρωπαϊκού προπολογισμού και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 17, της Ευρωζώνης. Με τα κονδύλια διάσωσης, το, τις ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 4,5% του ΑΕΠ, 3, με 4. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια διπλή ένωση. Αλλά οι ανώτερε κατηγορίε περιορίζονται σε 17 κράτη-μέλη. Δεν λέω ότι αυτό είναι κακό, αλλά τελικά εδώ βλέπουμε ότι ενώ προσπιζόμαστε την πολιτική συνοχή, αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα ουσιαστικά με την πολιτική συνοχή ήδη έχει διασωθεί μια πρώτη φορά. Επίση, είναι η δεύτερη φορά που θα πρέπει να αναφέρω την, το πόσο αγνώμη την εξωτερική διάσταση του προπολογισμού. Και αυτό είναι μια επένδυση. Ας μην ακολουθήσουμε την ε, κλασική στρατηγική του να βλέπουμε του εαυτού μα ω νησίδα ή νησί, όχι, βρισκόμαστε σε ένα διεθνέ προσκήνιο και από την άποψη τη εξωτερική δράση μπορεί να έχουμε και υλική επιστροφή και απόσβεση των επενδύσεων. Ασφάλεια, ε, σταθερότητα στην γειτονιά μα, ε, δημοκρατικά καθεστώτα, ε, αξίε και προβολή της δημοκρατίας. Τέτοιου είδους απόσβαση θα έχουμε μεταξύ του 2017 και 2012 η αύξηση στην εξωτερική δράση ήταν 30%. Τα επόμενα 7 χρόνια, το 2014, θα έχουμε επίπεδα χαμηλότερα από το 2013. Η αύξηση στα 7 χρόνια θα είναι 10%. Κανεί ε, ε, εδώ, παρόλο που μιλάμε για παγκόσμια Ευρώπη, για το διεθνέ προσκήνιο, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πολιτική είναι διαρθωτικά ε, και πραγματικά λιγότερο χρηματοδοτούμενη από ό,τι θα επιτρεπόταν. Η ασφάλεια είναι πιο σημαντική από την ευημερία. Η ε, στάθεια στη γειτονιά μα σημαίνει διακυμάνωση στι τιμέ των πετρελαίων, ανεργία, ε, μετανάστευση. Αυτά είναι πολύ σημαντικότερα από το 1% που προβλέπει ο, το, ο προπολογισμό. Η εξωτερική λοιπόν πολιτική θα έπρεπε να είναι κάτι που να προβλέπεται ω προτεραιότητα στον προπολογισμό, δημιουργεί ε, σταθερότητα, θέσει εργασία, ασφάλεια και δεν μπορεί να είναι παραμερισμένη. Θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα ενδιαφέροντά μα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Καρβάλιο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Υπουργοί, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία του να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ της του Ευρωπαϊκού και των υπόλοιπων ταμείων στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και στους εθνικούς. Είμαι εισηγήτρια για το ειδικό πρόγραμμα Horizon 2020, που όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε είναι το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία και την έρευνα στην Ευρώπη. Θα ήθελα εδώ να δώσω το παράδειγμα ακριβώς από το τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας όπου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπληρωματικότητα μεταξύ του Horizon 2020 και των διαφόρων εθνικών και περιφερειακών κονδυλίων και προγραμμάτων. Η φύση της, της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε σήμερα απαιτεί τις περισσότερες φορές ε, κρίσιμη μάζα, τη χρήση προηγμένων μέσων και κάτι που να λειτουργεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είναι τόσο περίπλοκη, περίπλοκη, περίπλοκη όρη της χρηματοδότησης ώστε θα πρέπει να εντείνουμε τις, προσπάθει, τις προσπάθειές μας για να έχουμε μια πολυτομιακή προσέγγιση και να γεφυρώσουμε τα χάσματα μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Για παράδειγμα, το Horizon 2020 θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα διαφορετικά ταμεία ώστε να επιτρέπεται η συμπληρωματικότητα και σχέση συνεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, από το Horizon 2020 θα μπορούσε να αντλούν ε, τα ταμεία της διάρθρωσης για την οικοδόμηση δυνατοτήτων και τη συμπληρωματικότητα. Αντιστρόφω, τα διαφορετικά ταμεία μπορούν να προλιάνουν το έδαφο από τι έννοιε τη γνώση προ τι ανάγκε τη αγορά, σηματοδοτώντα λόγου χάρη την επίδειξη τη πιλωτική φάση και να άρουν του φραγμού που μπορεί να εμποδίζουν του αγοραστέ. Νομίζω λοιπόν ότι τα διευθυντικά ταμεία στραμμένα προς την έρευνα και την καινοτομία θα μπορούσαν να συνδεθούν καλύτερα με προγράμματα όπως το Horizon 2020. Αλλά χρειαζόμαστε απλούς κανόνες για το σκοπό αυτό και ένα βαθμό συμβατότητα στους κανόνες συμμετοχής. Χρειαζόμαστε συντονισμό στην όλη διαδικασία της θέσης προτεραιοτήτων και στόχων. Άρα θα είναι ύψης της σημασίας να συνεργαστούμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που έχουν αναλάβει διάφοροι αρμόδιοι των ταμείων, μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των καθομελών πρέπει να αποφασίσουμε τις καλύτερες δυνατές πολιτικές και τα προγράμματα για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ακόμη τρεις, τρία μέλη που ζήτησαν το λόγο. Ε, παρόλο που τον πήραν ήδη σήμερα το πρωί. Θα τους δώσω το λόγο με την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μιλήσουν πάνω από ένα λεπτό. Ο κύριος ε, Σέτσικ από την Τσεχική Γερουσία. Ε, κύριε Πρόεδρε, πολλοί μίλησαν υποστηρίζοντας την ε, πολιτική συνοχή. Η Τσεχία θεωρεί ότι η πολιτική συνοχή είναι ιδιαίτερο σημαντική ε, στον πλαίσιο συζήτηση για τον προπολογισμό. Θα ήθελα να φέρω δύο πράγματα. Η γερουσία τη Τσεχία δεν επιθυμεί τη δημιουργία ενό αποθεματικού τη τάξη του 5%. Γιατί θα θεωρούσαμε ότι αυτό είναι μια, συνιστά μια ευκαιρία να τεθούν πιο χαμηλά οι στόχοι και κατά δεύτερο λόγο η αιρεσιμότητα ε, ενδεχομένως μπορεί να αποβεί προβληματική από την άποψη της επικουρικότητας. Η πολιτική της συνοχής είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο κατάχρησης. Ε, υποτίθεται ότι θέλει να ενισχύσει την ανάπτυξη σε ε, μειονεκτούσες περιοχές και όχι να οδηγήσει τελικά σε μια επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ο κύριος Κώστα Νέβες από την Πορτογαλική Βουλή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ένα λεπτό αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι Στηρίζουμε επί της ουσίας την προσέγγιση που έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτές τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Εν τω μεταξύ όμως βλέπουμε με κάποια σχετική ανησυχία τις ενδεχόμενες περικοπές στο πλαίσιο της ΚΑΠ, της πολιτικής συνοχής, πολιτικές που ούτως ή άλλως από τους στην πράξη υποστηρικτές τους δείχνουν ότι η συνοχή είναι απαραίτητη. Δεν είναι απλό απλώς ενδιαφέρουσα πολιτική, η πολιτική συνοχή, αλλά είναι και μια συνταγματική υποχρέωση. Προκύπτει από τις συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χώσε Μανουέλ Φερνάντες, εκ μέρους του ΕΛΚ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή ενίσχυσε μια πεποίθηση που είχα ευθύ εξ αρχής, ότι θα πρέπει να έχουμε μεθοδολογία αποτελεσματική για την κοινή αγροτική πολιτική και για την πολιτική συνοχή. Το Κοινοβούλιο ήδη το έχει πει ότι οι δύο αυτέ πολιτικέ δεν θα έπρεπε να γνωρίσουν περικοπέ στα κονδυλιά του. Όμω θα πρέπει να ξαναδούμε τα ποσά που διατίθεται στι δύο αυτέ πολιτικέ και εφόσον αυτά εξαντληθούν τότε να σκεφτούμε πώ θα χρηματοδοτηθούν άλλε πολιτικέ, άλλε προτεραιότητε, οι οποίε σωστά διερευνώνται στη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Η στρατηγική αυτή όμω ε, υπήρξε στο κέντρο των συζητήσεων διότι δεσμεύτηκαν τα κάτι μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο με πέντε στόχου που θα πρέπει να επιτευχθούν στο το 2020. Για να του πετύχουμε θα πρέπει τι επτά εμβληματικέ δράσει που έχουμε αναλάβει να τι φέρουμε ει εδώ όμως δεν είμαστε βέβαια για τη χρηματοδότηση. Επιπλέον χρειάζεται και μια άλλη προσέγγιση. Προσέγγιση bottom-up, από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή για την πολιτική συνοχή και την πολιτική την, και την ΚΑΠ χρειάζεται top-down προσέγγιση. Για τις υπόλοιπες bottom-up. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του πάνελ του δεύτερου γύρου των ομιλητών. Ένα τέταρτο για τις απαντήσεις, για τα σχόλια. Ε, θα ξεκινήσω με τον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Αυτή τη φορά ο κύριος Μπέγκε θα μας μιλήσει, συνεισηγητής για την έκθεση περί δημοσιονομικών προπτικών. Κύριε Μπέγκε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και βεβαίως θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα δείχνει τελικά ότι μόνο διορθωτικοί μηχανισμοί, εκτόσεις από τη μία πλευρά και δαπάνες που βασίζονται σε περισσότερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και στην ενίσχυση του πνεύματος της Ευρώπης 2020 ε, είναι αλληλένδετα ε, στοιχεία και δεν θα πρέπει ε, να το λησμονούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία θα πρέπει, και όλες οι συμφωνίες θα πρέπει να βασίζονται και στα δύο αυτά στοιχεία. Βεβαίω θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης, επικορικότητας και δημοσιονομικής πειθαρχία. Αυτό είναι απολύτω απαραίτητο. Προκειμένου να εξυγχρονίσουμε τον προπολογισμό, να κάνουμε σωστά πράγματα για την έρευνα και την καινοτομία, τι μελλοντικέ επενδύσει και για να συμπεριλάβουμε νέα δημοσιονομικά εργαλεία. Όλα αυτά είναι απολύτω αναγκαία. Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε την αλληλεγγύη και την ανάγκη ε, της ε, ενεργειακής ασφάλειας και ψηφιστικής ασφάλειας σαν μια βάση για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Και βεβαίως ε, θα ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά υπονομεύονται πράγματι από μια έλλειψη πραγματικής ευρωπαϊκής Συνεργασία. Θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ώστε να βρεθεί μια λύση μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου προκειμένου να αποφύγουμε καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των μελλοντικών κανόνων στο επίπεδο των χωρών μελών και επίσης καθυστερήσεις των πληρωμών όσον αφορά τα μεγάλα προγράμματα και τις ε, επενδύσεις που χρειάζονται οι χώρες και οι περιφέρειες. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι μια έκκληση προς την Δανική Προεδρία. Εκτιμώ πάρα πολύ πώς η διαδικασία που ξεκίνησε υπό την Πολωνική Προεδρία συνεχίζεται υπό την Δανική Προεδρία. Αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες οι συστάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα θέματα της διαπραγμάτευσης θα μέχρι τα τέλη του Ιωνίου και ε, οι συστάσεις μας να ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο και να μην παραμεληθούν. Δεν θα ήθελα να σας προειδοποιήσω, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι τα παραδείγματα όσον αφορά τις διαδικασίες συναπόφασης και όσον αφορά την προστασία δεδομένων, η απόρριψη της συμφωνίας αλίας με το Μαρόκο, ε, τέτοιες παραδείγματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι είναι καλύτερα να μιλούμε έγκαιρα μεταξύ μας παρά να κάνουμε ένα, μια μονόπλευρη συμφωνία και μετά να την ε, πετάμε στην κάλαθο των αχρήστων. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε ε, χρόνο, ότι χάνουμε χρόνο. Ε, μιλάμε για μια διαδικασία συναπόφασης στο, στο πολιτές δημοσιονομικό πρόγραμμα και καλό το Συμβούλιο να σεβαστεί αυτή τη διάκριση όσον αφορά τη συνένεση του Κοινοβουλίου. Το, χρειάζεται συνένεση του Κοινοβουλίου πριν πάρει ομόφωνα μία απόφαση το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την κατάθεσή του τα, ενώ τα πολιτή δημοσιονομικά προγράμματα βασίζονται στην διαδικασία της συναπόφασης. Και καλώ την Επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη της ως θεματοφύλακας της συνθήκης και να το κάνει αυτό απολύτως ε, ξεκάθαρα. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει μια συμφωνία για τις δαπάνες χωρίς μια πραγματική πρόοδο στους ιδίους πόρους. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο περιεχόμενο και το πνεύμα της συνθήκης, όχι μόνο εκεί που μας αρέσει και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το πούμε για ορισμένε χώρε που ανθίστανται στο περιεχόμενο τη συνθήκη. Σε σχέση με τα όσα είπε ο Ιταλό συνάδελφο ε, για την ευελιξία όσο πιο δύσκολα είναι τα στοιχεία, τόσο περισσότεροι η αριθμοί, ε, τόσο, μεγαλύτερη ευελιξία χρειάζεται στην ετήσια διαδικασία του προπολογισμού. Ε, το θέμα ε, του τι θα κάνουμε με τα μη δαπανηθέντα κονδύλια, ε, πώς θα μεταφερθούν στην επόμενη διαδικασία του προπολογισμού. Εδώ χρειάζεται αρκετή ευελιξία κάτι που δεν ε, συμβαίνει πάντοτε στις συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ξέρουμε, ε, ε, σήμερα το περισσότερο οι φίλοι της συνοχής και της αλίας εδώ παρόντες. Όχι τόσο εκείνοι που θέλουν να μειώσουν τις δαπάνες εκ μέρους του Συμβουλίου. Αλλά εγώ ξέρω πώς, πάνε, πώς γίνονται τα πράγματα στο Συμβούλιο. Ε, θα πρέπει να μιλούμε επίσης και για προσθέμενη αξία για απασχόληση και για ποιότητα των προγραμμάτων, καθώς και ε, κάποιων ε, προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ε, ανάγκες των χωρών μελών για την καταπολέμηση της ενεργείας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την απασχόληση. Λυπούμε που η Επιτροπή δεν απάντησε επαρκώς στην ανάγκη απλούστευσης των κανόνων ε, είτε στην, ε, όσον αφορά τη γεωργία, είτε όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Γιατί θα πρέπει εδώ να γίνει μια προσπάθεια προσαρμογή. Λέγεται ότι υπάρχει ένα επιπλέον γραφειοκρατικό άχθο τάξη 15-20%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις επιπτώσεις συνέργειας, τα αποτελέσματα συνέργειας μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικών προπολογισμών. Και αυτή η συνδιάσκεψη, η συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι οι πρόεδροι των κοινοβουλίων θα πρέπει ε, να βρουν ε, κάποιες ευκαιρίες, ε, κάποιες ημερομηνίες στον προγραμματισμό τους ούτως ώστε να γίνονται τέτοιου είδους συναντήσεις γιατί συνιστούν μια καλή ευκαιρία για να δημιουργεί ένα σωστός ευρωπαϊκός ε, δημόσιος διάλογος ε, στον οποίο να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι τίποτε δεν ε, μπορεί να συμφωνηθεί αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλες οι λεπτομέρειες. Οι οροφές για το 2013, για το MFF, ε, θα παραμείνουν ως έχουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει να μειωθούν αυτοί οι αριθμοί, αυτά τα ποσά. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Βάιτ από το Ελλανδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πρόεδρε ε, συνόψισε πολύ καλά την σημερινή συζήτηση και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η σύνοψή του, αλλά κύριε Πρόεδρε για μένα ήταν πολύ πλούσια η συζήτηση αυτή. Ε, κέρδισα πολλά από αυτήν η φιλοδοξία για την οποία μιλούσαμε νωρίτερα. Πιστεύω ότι υπάρχει. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να σκεφτούμε πώς μπορεί αυτή η φιλοδοξία να πραγματοποιηθεί ...εάν ακολουθήσουμε τις περικοπές στον προϋπολογισμό. Τα γεγονότα δείχνουν ότι αν η φιλοδοξία που ακούσαμε σήμερα θέλουμε να πραγματοποιηθεί, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για περικοπές στον προϋπολογισμό. Και εγώ πρόσεξα ότι ακούσαμε διάφορες φωνές που ήθελαν ε, λιγότερες ε, δαπάνες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, όπως είπε ο κύριος Πέκε, ότι πρέπει να ε, συμπληρώσουμε και την άλλη μεριά της εξίσωσης. Θα πρέπει να πάμε στις, κοινων... στις διάφορες κοινωνίες, στους ψηφοφόρους μας, στους μας να ε, τους εξηγήσουμε όχι μόνο ε, πώ έχει η κατάσταση, αλλά να του ε, δείξουμε ότι χρειαζόμαστε τι δαπάνε αυτέ. Ε, πρέπει να το εξηγήσουμε σε αυτού, διότι αυτοί ε, λαμβάνουν αποφάσει ουσιαστικά με, τις, με του φόρου που συνεισφέρουν. Και κύριε Πρόεδρε, δύο τελευταία πράγματα που θέλω να τονίσω από σήμερα. Άκουσα την ισορροπία που πρέπει να διατηρήσουμε ανάμεσα στη δίαιτα και τον αθλητισμό. Το εκτιμώ πολύ αυτό. Ε, ίσως εγώ προσωπικά να μην κάνω πολύ δίαιτα, αλλά η χώρα μου ε, κάνει πολύ δίαιτα, ίσως δεν αθλείται αρκετά. Αν έχουμε λοιπόν μια πολιτική που συνδυάζει και τα δύο, μπορεί να χρειαζόμαστε λιγότερη δίαιτα, πιο νωρί από ό,τι πιστεύαμε. Και η τελευταία έννοια που συγκρατώ από τη συζήτηση αυτή είναι η έννοια της αλληλεγγύης ε, και νομίζω ότι αυτό ε, υπήρξε σε πολλές παρεμβάσεις που ακούσαμε και αυτό είναι συγκινητικό. Ε, ε πολλοί ομιλητές μίλησαν για την ανάγκη να διατηρήσουμε τα ταμεία συνοχής ε, και το τόνισαν αυτό. Οι φωνές αυτές ε, που μιλάνε για την διατήρηση των ταμείων συνοχής πρέπει να ακουστούν. Και τέλος και κύριε Πρόεδρε, Πρέπει να συγχαρούμε τη Δανέζικη Προεδρία για τη δουλειά που έχει κάνει και σήμερα και που πραγματοποιείται σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Κυπριακή Προεδρία θα αναλάβει τα ενία στα μέσα της χρονιάς και αν ε, ολοκληρωθεί ο στόχος μέχρι το τέλος της χρονιάς όπως ε, ελπίζουν πολλοί, ε, πιστεύω ότι θα υπάρχει αρκετή δουλειά που θα απομένει να γίνει για την επόμενη Προεδρία που είναι η Ιρλανδική Προεδρία που θα αναλάβει τα ενία στην αρχή τη επόμενη χρονιά. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε να συζητήσω εδώ σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και είμαι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε. Σας ευχαριστώ κύριε White, κυρία Κρού. Ελέγχθησαν πολλά σε σχέση με την συνοχή. Ωστόσο υπάρχει μια συνοχή μεταξύ του Horizon 2020 ε, της ε, διασύνδεσης και ε, ένα σημαντικό θέμα είναι η καινοτομία και η έρευνα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ωστόσο, ε, η συνοχή μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερο ουσιαστική γιατί θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους. Για να το πούμε με καθημερινούς όρους, εάν τους διασυνδέσουμε με το σωστό τρόπο θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους, οι επιπτώσει τους. Τώρα, όσον αφορά με μη δαπανηθέντα κονδύλια, ε, είχα μια, μια σχετική εμπειρία στην προηγούμενη επιτροπή σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο. Εκεί υπήρχαν τέτοια χρήματα που δεν είχαν ταπανηθεί και λήφθη η απόφαση και η οποία έγινε αποδεκτή από όλου να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό για αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν χρήματα που συναντούσαν με ένα φλιτζάνι καφέ, αλλά 100 ε, εκατομμύρια ευρώ. Και ε, τελικά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό γιατί οι χώρες μέλη αποφάσισαν να πράξουν διαφορετικά. Και ήθελα να πω αυτό προς τον Ιλανδό, Ολλανδό εκπρόσωπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μείωση τουλάχιστον του 5%. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα και νομίζω ότι ε, μόνο τα παραδείγματα είναι καλά να μας φωτά το πνεύμα των μεγάλων συνδιασκέψεων. Όταν μιλούμε για την έρευνα και την επιστήμη, θα ήθελα να πω ότι ε, τη διάρκεια αυτού του πάνελ ε, θα έχουν δημοσιευθεί 500 καινούρια επιστημονικά άφρα. Θα έχουν δει το φως στις δημοσιότητες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τους επιστήμονες και τους φοιτές μας ότι έχουν την επαρκή πρόσβαση σε αυτά τα επιστημονικά άφρα. Έχουμε ανάγκη νέων εργαλείων ε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτή η νέα καινοτόμο προσέγγιση για την κοινωνία μας και την οικονομία μας. Και Έχουμε ήδη ένα υψηλής ταχύτητας ε, διαδίκτυο το οποίο διασυνδέει τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρώπης. Πάνω από χίλιες φορές ε, ταχύτερο από, τα, από τις ευρυζωνικές μας ε, υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του, της Ευρώπης 2020. Και πραγματικά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, συνεργασία λοιπόν μεγάλης ε, κλίμακας ε, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Και ένα τελευταίο παράδειγμα όσον αφορά την ε, ενημέρωση για την υγεία. Και ε, αν εξετάσουμε τα μεμονωμένα μας συστήματα θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα περί υγείας και να φτάσουν στους ασθενείς θα πρέπει να υπάρξει επαρκής, καλή συνεργασία όσον αφορά αξιόπιστες ε, στατιστικές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της υγείας και να δώσει μια κινητήρια δύναμη θα πρέπει είναι συμβατό βεβαίω με τι ε, προτάσει για την μεταρρύθμιση όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ψηφιακά συστήματα υψηλή ε, ταχύτητα. Και αυτά όλα εννοώ με το Interconnect Europe. Ε, παρακαλώ να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σα, γιατί πραγματικά αυτά είναι το μέλλον μα και το μέλλον μα ξεκινάει αυτό το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νικολάη ε, Ταυκυλιέβιτς από το, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας. Um, Δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο, την Προεδρία, την Επιτροπή που διοργάνωσαν αυτήν την ε, διάσκεψη. Νομίζω ότι εκπληρώσαμε ένα πολύ σοβαρό καθήκον. Είμαστε σε πολύ ενδιαφέρον στάδιο στις διαπραγματεύσεις. Ακόμη και αν δεν ξέρουμε εάν θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ή όχι. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε εν τέλει ω προς το περιεχόμενο. Ξέρουμε όμως ότι έρχεται μια καμπή πολύ σύντομα. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση σήμερα με όλες τις ε, συνεισφορές και τις ανταλλαγές απόψεων που είχαμε, ιδίως με την παρουσία των κάτω μελών και του Συμβουλίου, που άκουσαν διαφορετικές ε, τοποθετήσεις. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλό που οι υπέρμαχοι τη συνοχή ε, κινητοποιήθηκαν σήμερα. Δείχνει αυτό ότι πραγματικά είμαστε και συνεκτικοί και δραστηροί. Όμως είμαστε ελαφρώς ε, ε που οι φίλοι μας από τα κράτη πληρωτέ ήταν πιο σιωπηλοί. Τι σημαίνει αυτό. Δεν τους έψαν τα επιχειρήματα. Ελπίζω όχι. Και χωρί να είμαι αφελή, θα έλεγα ότι ο λόγο είναι ότι ίσως θέλουν τους μεγάλους αριθμούς να τους συζητήσουν σε άλλη φάση, σε κατοπινό στάδιο, όταν θα είναι τα πράγματα κρίσιμα και θα πλησιάζει η στιγμή της λήψης αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση θέλω να στηρίξω την ιδέα που είναι προσφυλής και στην Δανική Προεδρία ότι πρέπει όντω αυτή η συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είναι όσο δυνατόν διαφανέστερη. Ήταν πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία σήμερα. Second uh, is uh, that... Το δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε διαφορετικέ απόψει. Νομίζω η συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετατοπίστηκε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το τελευταίο εξάμεινο σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Όλοι παραδέχονται σήμερα ότι η ανάπτυξη, οι επενδύσει, οι νέε ευκαιρίε, η ανταγωνιστικότητα είναι πυλώνε του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, διότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβλήθηκε με, με τι καλύτερε δυνατέ προποθέσει και ήταν καλή, αλλά όχι τέλεια. Τώρα νομίζω ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη. Θυμάμαι πολύ καλά τον Ιούνιο πέρσι, οι συζητήσεις περισσότερο αφορούσαν το τι γίνεται με το χρέος, τη δημοσιονομική εξυγίανση σε αντίθεση με τις δαπάνες. Είναι ενθαρρυντικό που σήμερα έχουμε πάρει πια μια ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση. Τουλάχιστον με αφορμή το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερος και ανυπομονώ για την επόμενη διάσκεψή μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Euh, Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση του δεύτερου γύρου τραπέζης της ε, ημερίδας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο εξυπηρετικοί ώστε να μπορέσω να διευθύνω σωστά τι συζητήσει σε αυτού του δύο γύρου. Με τέσσερα λεπτά μόλι σεβαστικά με το χρόνο μα κατά τα άλλα, περνάμε στα συμπεράσματα τη ε, ημερίδα. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την Προεδρία να αναλάβει ο κ. Σεύκοβιτ, Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Λαμασούρ, Πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ο Υπουργό Βάμεν, ε, υπεύθυνο για ευρωπαϊκέ υποθέσει από το Δανικό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ όλου. Μπορεί να δουλεύαμε όλη τη μέρα, αλλά ακόμη μας έχει μείνει κάμπος η δουλειά. Με ιδιαίτερη χαρά, καταλαμβάνω τη θέση αυτή, με δύο φίλους κοντά μου. Ο πρώτος είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μάρος Σεύκοβιτς, και ο άλλος είναι μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Αλά Λαμασούρ. We would now θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω τις εντυπώσει μας σε σχέση με τι διαπραγματεύσεις για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο και το τι έχουμε να συναντήσουμε μπροστά μας. Είναι σαφέ το μήνυμα. Είμαστε εδώ καθισμένοι χαμογελώντα. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, όλοι μαζί. Άρα, η μέρα είναι μπροστά μας. Χωρίς λοιπόν επιπλέον καθυστερήσεις να δώσω το λόγο στον κύριο Λαμασούρ, τον οποίο θα ήθελα και να συστήσω, να τον παρουσιάσω λέγοντας ότι είναι από τα εμπειρότερα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά είναι και από τους ε, ανθρώπους που όταν διορίστηκα υπεύθυνο των ευρωπαϊκών υποθέσεων ένας από τους πρώτους που μίλησε ήταν ο κύριος Λαμασούρ ξεκινήσαμε όμω με τι διασκέψει αυτού του τύπου επί πολωνική προεδρία. Γι' αυτό σα έστηκε πολύ πρόσφατο στη θέση αυτή και σε αυτή την ε, ιδιότητα. Είσαστε ο πατέρα τη ιδέα αυτών των ημερίδων. Κύριε Λαμασούρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νικολά, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ανική Προεδρία που διοργάνωσε από κοινού με το Κοινοβούλιο, με τον Πρόεδρο κύριο Σούλτς, αυτή τη διάσκεψη, μετά την Πολωνική διάσκεψη και έχοντας αντλήσει τα διδάγματα από την Πολωνική διάσκεψη και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβούλων που ήρθαν από μακριά και συμμετείχαν στο σύνολο των εργασιών. Ε, διαπίστωσα ότι μεταξύ των 27 που τώρα είναι, σήμερα, που τώρα είναι 28 συν την ε, Κροατία, 11 ήταν, εκπροσωπούνταν σε υπουργικό επίπεδο, 20 από βουλευτές, και αυτό το οποίο με εντυπωσίασε σε σύγκριση με την πρώτη συνάντηση είναι το γεγονός ότι ε, τώρα πλέον αρχίζουμε μία αληθινή ανταλλαγή απόψεων. Όχι μία διαπραγμάτευση, γιατί αυτή γίνεται σε ένα άλλο πλαίσιο, αλλά μία ανταλλαγή της, ε, των εις αναλύσεων. Η κρίση αποκάλυψε πολλά πράγματα και σε όλες τις χώρες, σε όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσπούνται εδώ, ε, μοιραζόμαστε τον διτό στόχο, την εξηγήνση του προπολογισμού και την ε, ενίσχυση της ανάκαμψης. Και εδώ βλέπουμε το μέλλον της Ευρώπης. Όσον αφορά τους φόρους σήμερα το πρωί, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, παρόλο που βεβαίω υπάρχουν και αποκλήσεις όσον αφορά τις λύσεις που προτείνονται. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το υφεστάμενο σύστημα των πόρων που τροφοδοτούν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, σύστημα που θεσπίστηκε πριν από 20 χρόνια, δεν λειτουργεί πλέον και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Πολλά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων επέμειναν ε, στο θέμα της ε, δημοσιονομικής ε, κυριαρχίας των χωρών μελών. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν διακυβεύεται. Δεν τίθεται να αμφιβόλο. Οι προτάσεις που είναι στο τραπέζι αποβλέπουν σε ένα σύστημα ιδίων πόρων, έτσι όπως προβλέπεται από τη συνθήκη και εγγράφεται στη συνθήκη και λειτουργήσε τα πρώτα 30 χρόνια και με ένα συγκρίσιμο τρόπο με το σύστημα από το οποίο αποφελούνται πολλές ε, περιφέρειες και πόλεις. Δεν πρόκειται για ένα θέμα μεταφοράς της κυριαρχίας εδώ. Δεύτερον, θα ήθελα να επιμείνω όσον αφορά τους πόρους, ότι αν συμφωνήσουμε για να δημιουργήσουμε νέους ιδίους πόρους ή να να πρικοδοτήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, το σύνολο των ιδίων πόρων θα ε, μειώσουν πράγματι τις εθνικές δαπάνες, είτε άμεσα αν ένα τμήμα αυτών των πόρων, για παράδειγμα, να φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών διατηρηθεί από τις χώρες μέλη, είτε έμεσα, γιατί τα δύο τρίτα που θα τροφοδοτήσουν την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό θα εκπέσουν από την εθνική εισφορά των χωρών μελών. Άρα ε, εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα στο 100% για τις χώρες μέλη. Όσον αφορά τώρα τις δαπάνες, νομίζω ότι όλοι ε, κατανόησαν ότι σήμερα έχουμε 27 εθνικού προπολογισμού, σύντομα θα έχουμε 28 και ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι ο 29ο. Είναι ο κοινό προπολογισμό τη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ούτως ώστε να ανταποκρίνεται βέλτιστα στις σημερινές ανάγκες και βλέπουμε, όπως είπε ο Άλεξ Βάιτ, εξ ονόματος του Ελλανδικού Κοινοβουλίου, ότι η υποστήριξη της οικονομικής ε, μεγέθυνσης την οποία χρειαζόμαστε, δεν μπορεί να γίνει σήμερα με απολυσματικό τρόπο, παρά μόνο στο πλαίσιο των 27, ε, χρησιμοποιώντας, εξοπλώντας τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η μεγάλη κίνδυνη, τη οποία ανέφερα χθε στο δείπνο, ε, η μεγάλη κίνδυνη που θα πρέπει είπατε, να αποφύγουμε είναι να ξαναβρεθούμε το 2020 με έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό, του οποίου ε, το ποσό, η προτεραιότητα, η δομή και η χρηματοδότηση θα είναι ακριβώς ε, αυτή του προπολογισμού του 1990. Αυτό δεν είναι πλέον δυνατό. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια ε, κοινή γεωργική πολιτική το 2010 ή το 2020 από αυτή που ανταποκρινόταν στις ε, ανάγκες του 2000. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένε χώρες δυστυχώ διασπαθίζονται οι πιστώσει, ενώ ε, και σε άλλε χώρες δεν ήξεραν να δαπανίσουν τα κονδύλια, δεν αποφευθήθηκαν δηλαδή, άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και όσον αφορά την πολιτική της έρευνας υπόθηκαν πολλά σημαντικά πράγματα. Όσον αφορά την ενεργική πολιτική, στο εξή ε, η Ένωση έχει μια αρμοδιότητα. Δεν είναι δυνατόν να βρούμε σαν να μην υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε καταλήλω την ευρωπαϊκή πολιτική και να την προκοδοτήσουμε με τα μέσα. Τέλος, έχουμε ανάγκη ευελιξίας. Έχουμε το πλεονέκτημα να πλαισιώνουμε τον προπολογισμό, να τον καταρτήσουμε για μια περίοδο 7 ετών υπάρχει βεβαίω ένα ε, ε, κίνδυνο ακαμψία, γιατί υπάρχουν κάποιες απρόβλεπτε εξελίξει. Όταν θέλησαμε να προσαρμόσουμε για παράδειγμα το πλάνο ανάκαμψη για να καταπολεμήσουμε την ύφεση ε, χρειάστηκαν να πολλά χρόνια ή όταν οι γαλακτοπαραγωγοί έχασαν 30% των εσόδων του. δεν μπορέσαμε να του βοηθήσουμε. Όταν οι χωρικοί της Αφρικής ήταν θύματα της αύξησης τη τιμή των σπόρων και των ε, χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια σε ότι οι Αφρικανοί ε, καλλιεργητές επωφελθούν τις πρώτες ενίσχυσης εκ μέρους του Μπαρόζο. Ε, λοιπόν, πιστεύω κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν ε, στο να εμπλουτίσουν το negotiating box, ε, το πακέτο της διαπραγμάτευσης για την Δανική Προεδρία και νομίζω ότι θα πρέπει να ανανεώνουμε ε, τέτοιου είδους συζητήσεις βάσει ενός χρονοδιαγράμματος βεβαίως, ούτε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια σύμπλευση των κοινοβουλευτών των βουλευτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλέν, για αυτήν την τόσο στρατευμένη σου παρέμβαση, ο κ. Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ, Νικολάη, ε, αλλά βουλευτές, ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Ευρωκοινοβούλιο και την Τανική Προεδρία που φιλοξένησαν αυτήν την δεύτερη συνδιάσκεψη. όπω μόλι υπόθηκε, ο Αλά είναι πατέρα αυτή τη ιδέα, αλλά ο Νικολάη ήταν ε, ο πρωτεργάτη της δεύτερης αυτής ημερίδα, ώστε να οργανωθεί μάλιστα εδώ στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν συνέχεια στι όλε τι συζητήσεις για τα τόσο σοβαρά ζητήματα που μα απασχολούν για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε επισκέπτες και από τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ. Όπως γνωρίζετε, συχνά συζητώ με τα Εθνικά Κοινοβούλια και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τέτοια ειδικά φόρα για την ανταλλαγή απόψεων. Είναι μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε οι μεν τις απόψεις των ΔΕ, να δούμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα από διαφορετικές σκοπιές και να καταλάβουμε ή μεν την αντίληψη των δε. Είναι λοιπόν πολύ καλή ευκαιρία να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να έχουμε εκπροσώπους από όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι μεγάλη ικανοποίησή μου γιατί υπήρξε ενεργή συμμετοχή από την Επιτροπή των Περιφερειών και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Και οι δικές τους απόψεις έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών των κρατών Οπότε θα πρέπει με άκρα προσοχή να αφουγκραστούμε τις απόψεις και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρώπης, αλλά και των δύο Ευρωπαϊκών Επιτροπών. Επίσης, να υπογραμμίσω το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν θα είναι αρκετά δυσχερείς. Οπωσδήποτε δεν θα είναι απλό να επιλέξουμε τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τις προσθεσμίες τους ερχόμενους μήνες. Θα χρειαστεί σκληρή, εντατική δουλειά από όσους έχουμε μπλακεί στην όλη διαδικασία και νομίζω ότι για αυτό το λόγο θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε αυστηροί στον ορισμό των κονδυλίων θα χρειαστεί για την επόμενη περίοδο δαπανών, για το επόμενο πολιετέ πλαίσιο κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Είδαμε τι απόψει ε, διαμορφώνονται για το τόσο σοβαρό ζήτημα αυτό. Και όπως ακούσαμε από πολλές παρεμβάσεις, δεν μπορούμε να γνώμε το σημερινό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τοπίο. Ε, Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να δώσει τα απαιτούμενα αποτελέσματα και να στηρίξει τις ε, κοινώ συμφωνημένες πολιτικές μας ε, με τις κατάλληλες επενδύσεις τις, στους σωστούς τομείς. Νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να πούμε ότι είχαμε μια επικοδομητική, μια πλούσια συνδιάσκεψη που μας επέτρεψε να δαπανίσουμε με τρόπο ορθό το χρόνο που μας διατέθηκε για τις δαπάνες και τους στόχους του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Στην εισαγωγή του σήμερα ο πρόεδρος Μπαρόζο έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην προστιθέμενη αξία των δαπανών του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε σχέση με αυτές των εθνικών προπολογισμών. Εγώ άκουσα την στάση που εξέφρασε η κυρία Κρούς, όπου στο προηγούμενο γύρο ομιλητών έδωσε πολύ σαφή παραδείγματα αυτού του γεγονότος. Το στοιχείο αυτό προέκυψε και από τις συζητήσει μου με τα εθνικά κοινοβούλια. Διότι όταν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε σύγκριση με τους εθνικούς πρέπει να δούμε ότι είναι σαφής η ανάγκη να υπάρχει πραγματική αξία. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό πρέπει να προσφέρει κάτι και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Επίτροπο Λεβαντόφσκι, στην πρώτο κύριο Μιλητών, μα είπε ποια θα είναι η προσέγγιση τη Επιτροπή ω προ του πόρου. Όπω όλοι ακούσατε, η Επιτροπή καθοδηγείται από το να αντικαταστήσει την παρούσα κατάσταση και τους κανόνες που θεωρούνται περίπλοκη από ένα σύστημα απλούστερο, διαφανέστερο και συνδεδεμένο με τους πολιτικούς στόχους. Εξήγησε ο κ. Λεβαντόφσκι πως γενικός ο φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση κατά 50% τουλάχιστον του, της συνεισφοράς του ΑΕΠ των 100 μελών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν δύο τρίτα διατίθενταν από αυτό το φόρο, θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι ήδη πόροι. Η θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα τονίζει την ανάγκη να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση ω προ τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω ότι σε όλου, ε, από τις παρεμβάσεις όλων αποδόθηκε προσοχή στο γεγονός αυτό. Η ίδια συνδιάσκεψη το αποδεικνύει. Ο ίδιος ο πρόεδρος Σούλτ το είπε. Η Σημασία του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου γνωρίζετε και από τη Δανική Προεδρία τι προσεχεί εβδομάδε και μήνε. Θα πρέπει να αντιδικοποιήσουμε τη συνεργασία μα προκειμένου με τους βασικούς φορείς όπως τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον ε, Χέρμαν Φαρόμποη, να προωθήσουμε την όλη διαδικασία. Εάν ε, παραπέμψω σε άλλες φάσεις της συζητήσης, Νομίζω ότι παρόλα αυτά θα δούμε ότι υπήρξε συνένεση για το ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός είναι εργαλείο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και ο προπολογισμό αυτός μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, συμφωνούμε ότι η λιτότητα είναι απαραίτητη και πρέπει οι δημόσιες δαπάνες μας να εξηγιανθούν. Όμω τα μέτρα λιτότητα πρέπει να συνοδεύονται από επενδύσει στι υποδομέ, στην έρευνα, στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τα μέτρα που θέλουν να ευνοήσουν την ανάπτυξη. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό θα είναι ένα καθοριστικό αποτέλεσμα τη στρατηγική για την Ευρώπη το 2020. Με χαρά θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις που έγιναν από πολλούς ομιλητές σήμερα γύρω από το γεγονός ότι η συνοχή θα παραμείνει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να καλυφθούν οι ανισότητε και αποκλήσει μεταξύ των κατομελών και στο ερχόμενο χρονικό διάστημα. Εκπρόσωποι των νέων κατομελών, αλλά όχι μόνο από τα νεα κάτι κράτη-μέλη, ζήτησαν την ε, συνέχεια επίδειξη αλληλεγγύη μέσω των κονδυλίων τη πολιτική συνοχή και των διαθετικών ταμείων. Υπάρχουν βέβαια και διαφωνίε και μπορούμε να πούμε ότι οι απόψεις ε, αντιφάσκουν σε κάποια στοιχεία της πολιτικής αυτής, όπως η θέση ορίων ή τα αποθέματα για τις επιδόσεις, ε, η ανταμοιβή των επιδόσεων, κάτι που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Όμως νομίζω όλοι συμφωνούμε στο εξή. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν αφορά μόνο τα ποσά, τα αριθμητικά ποσά, αλλά είναι ένας τρόπος να ορίσουμε το επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Είναι ένα σαφές μήνυμα για το τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να δημιουργήσουμε για το μέλλον. Και Νομίζω ότι η ερώτηση αυτή είναι περισσότερο εύστοχη όταν συζητάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις στιγμές κρίσης. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε με αυτό το μήνυμα από τη διάσκεψη. Δεν θα είναι απλέ οι διαπραγματεύσει για τα αριθμητικά ποσά. Ότι όλοι θέλουμε να ελπίζουμε ότι η δανική Προεδρία θα το διευκολύνει όλα αυτά, το ίδιο και το Συμβούλιο, και ότι όλοι μαζί θα βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ των επενδύσεων, τη αλληλεγγύη και των φιλοδοξιών μας. Νομίζω ότι απότερος στόχος μας θα πρέπει να είναι να επιτύχουμε συμφωνία, τελική συμφωνία μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ώστε να βεβαιωθούμε ότι το 2014 ο ετήσιος προπολογισμός θα είναι έτοιμος εγκαίρος και τα ανάλογα προγράμματα και εργαλεία θα αρχίσουν να λειτουργούν από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Η Ευρώπη χρειάζεται πλέον ε, θετικές ειδήσει. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση και βλέπουμε ότι χρειάζεται ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι υπάρχει κάποια απόφαση για την ανάπτυξη, για τον προπολογισμό που θα ευνοεί την ανάπτυξη. Ω το 2020 Κάτι τέτοιο θα ήταν μια σαφή ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σκληρά για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τη, ότι επιδεικνύει αλληλεγγύη και ότι ετοιμάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόσμο του 21ου αιώνα. Συμπερασματικά, ήθελα να πω ότι το καθήκον μα δεν θα είναι απλό. Πιστεύω ακόμα ότι είμαστε στη σωστή τροχιά για να καταλήξουμε σε συμφωνία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο τέλος της χρονιάς και αυτή η συμφωνία θα πρέπει να εξισορροπήσει μεταξύ φιλοδοξιών και στόχων τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι το χρωστάμε στου Ευρωπαίου πολίτε, το χρωστάμε στου εταίρου και θα πρέπει να αναζητήσουμε ακριβώ του τρόπου που θα φέρουν προς τη θεμένη αξία και εξυγχρονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Ο Νικολάη ξεκίνησε το γύρο αυτό λέγοντας ότι υπάρχει αισιοδοξία στην αίθουσα και ότι ήδη χαμογελάμε. Όχι μόνο εμείς, πολλοί και από τους ευρωβουλευτές. Και κατά κύριο λόγο και ο κύριος Μπέγκε χαμογελούσε. Αυτό είναι σαφής ένδειξη, σαφής ένδειξη ότι κάτι καλό κάνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, για την ενεργό του συμμετοχή και το Ευρωκοινοβούλιο και τη Δανική Προεδρία για τη διοργάνωση αυτής της ε, διάσκεψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, για την πολύ καλή ομιλία σας και σας ευχαριστώ που μοιράζεστε και την αισιοδοξία του κυρίου Πέγκο και άλλων εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές. Κάποιες χώρες θα ήθελα ο προπολογισμό να παραμείνει ως έχει ή να αυξηθεί. Άλλοι θα θέλανε μείωση του προϋπολογισμού. Μερικά κράτη-μέλη θα προτιμούσαν να δώσουμε πολύ προσοχή στην κοινή γεωργική πολιτική, άλλοι στην πολιτική συνοχής. Αυτό που μας ενώνει όμως, εδώ σε τούτη την αίθουσα, είτε προερχόμαστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ή κοινοβούλια των κρατών μελών είναι η σαφής υποχρέωση να καθορίσουμε την πορεία για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Καθορίζοντας έτσι και την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να μετακινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 500.000 εκατομμύρια πολίτες που περιμένουν να συνεργαστούμε. Η Ευρώπη βρίσκεται στην βαθύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε κάνει πολλά απαραίτητα βήματα για να σφίξουμε το ζωνάρι με μέτρα λιτότητας. Και αρχίζουμε να βλέπουμε το φως στο τέλος του τούνελ. Δεν θα το πετύχουμε αυτό όμως εάν ε, τα θεσμικά όργανα ε, μάχονται μεταξύ τους. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο με τη συνεργασία. Γι' αυτό η Δανέζικη Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τους επόμενους μήνες να προωθήσει το θεματολόγιο όσο γίνεται ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό αυτού του χρόνου, να μπορεί να ε, ολοκληρωθεί το θέμα και να επιτευχθεί συμφωνία. Αυτό θέλει η Ευρώπη. Θα επενδύσουμε στην ανάπτυξη, θα επενδύσουμε στην απασχόληση για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή 23 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εκατομμύρια νέους οι οποίοι μας κοιτούν σήμερα και ζητάνε λύσεις. Ζητούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, όποια και αν είναι η ευθύνη μας, σίγουρα συμμεριζόμαστε αυτήν ε, την υποχρέωση. Θα ήθελα εκ μέρους της, Ευρωπαϊκ... της να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, για την πολύ στενή συνεργασία, όχι μόνο κατά την διοργάνωση αυτής της διάσκεψης. Και όπως είπε ο Αλέ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη. Δύο πατέρες έχουμε. Εγώ θα έλεγα ότι ένας είναι ο πατέρας εδώ. Ε, πάντως, ε, χάρηκα που μπόρεσα να βοηθήσω. Συναντιόμαστε όμως τακτικά πριν από κάθε ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όπου συζητείται το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φτάνει στο τραπέζι των Υπουργών. Ακούγεται η φωνή σας λοιπόν. Ελπίζω ότι και εσείς από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχετε στενή συνεργασία με τις δικές σας κυβερνήσεις από όπου και αν προέρχεστε. Διότι Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Κάθε 7 χρόνια έχουμε την ευκαιρία αυτή. Δεν θα υπάρχει λοιπόν δικαιολογία εάν αποτύχουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσά που ε, μας δώσατε το χρόνο σας. Έχετε ε, πολλή δουλειά στις πατρίδες σας. Και σας υπόσχομαι όχι ότι κάθε δήλωση θα ε, μετατραπεί σε χρήματα στον προϋπολογισμό, κάθε δήλωση όμως ε, θα, θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στην ε, διαδικασία που μας περιμένει. Και είμαι πεπισμένος ότι αν συνεργαστούμε θα είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνία στο δεύτερο μέρος της φετινής χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Λήξη τη συνεδρίασης. Thank